Good morning, and gentlemen. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρακαλώ καθίστε. Για να ξεκινήσουμε την πρωινή μας συνεδρίαση της Επιτροπής Ρέτζι. Ευχαριστώ. να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις 24 25 Ιανουαρίου. Το σημείο αυτό είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης της έκθεσης της Επιτροπής ΕΚΟΝ με θέμα το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντανισμό των Οικονομικών Πολιτικών ετήσια έκθεση ανάπτυξης 2018. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένας ετήσιος κύκλος οικονομικής και δημοσιονομικής ε, πολιτικής και συντονισμού αυτών μεταξύ των κρατών μελών. Επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της να συζητήσουν τον προγραμματισμό τους για την οικονομία και τον προπολογισμό και να παρακολουθήσουν την πρόοδο σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στο έτος. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ έχει αξιοποιήσει δύο, ε, ε, μάλλον συντάσσει δύο εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας ετησίω ε, για τη δικασία αυτή, μία την Άνοιξη και μία το Φθινόπωρο. Η έκθεση τη άνοιξη βασίζεται στην ετήσια έκθεση ανάπτυξη τη Επιτροπή για την επόμενη χρονιά και είναι μία απόπειρα να επηρεαστούν οι ετήσιε οικονομικέ και κοινωνικέ προτεραιότητε που εγκρίνονται από, το ερεινό, από την Ερεινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ συνέταξε τώρα την έκθεσή της της Άνοιξης για το 2018 βασιζόμενη στις προβλέψεις για τη χρονιά αυτή που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως δημοσιεύτηκε στις 22 Νοεμβρίου του 2017. Η Επιτροπή ζητά από την Πρόεδρο να συντάξει γνωμοδότηση εκ μέρου τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη και αυτή θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα. Λόγω του χρονοδιαγράμματο τη καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή ΕΚΟΝ θα πρέπει να ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μα του Φεβρουαρίου. Γι' αυτό προτείνω μια σχετικά σύντομη προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών στο τέλος της εργάσιμης ημέρας 3η 30 Ιανουαρίου 2018 στις 5 το απόγευμα. Θα παρουσιάσω τώρα το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Και μετά θα συζητήσουμε με τους κοιόδης εισηγητές και τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζι. Και τώρα θα μιλήσω τη βουλγαρική γλώσσα. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, έχω την χαρά να σας παρουσιάσω την ε, θέση της δικής μας Επιτροπής ε, για ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της σχετικής διαδικασίας. Πρόκειται λοιπόν ε, για μια γνωμοδότηση όπου αναφέρουμε ότι φαίνεται να δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψη η οικονομία στην Ευρώπη. Έχουν κάποια θετικά στοιχεία, χαμηλά ποσοστά ανεργία, τα χαμηλότερα από τότε που ξέσπασε η κρίση. Βέβαια, αναφέρουμε ότι αυτή η ανάκαμψη δεν ε, φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα σε όλα τα κράτη-μέλη, γιατί σε πολλέ περιφέρειε τη Ευρώπη η ανεργία είναι πολύ υψηλή ιδίω η νεανική ανεργία. Και λέμε ότι πρέπει να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο τη συνοχή και τη σύγκληση και τη θετικής δυναμικής που φαίνεται να επιβεβαιώνεται σε σχέση με την ανάκαμψη στην Ευρώπη. Υπάρχουν οι συστάσεις χώρα, αλλά βλέπουμε ότι δεν προχωρεί η εφαρμογή των συστάσεων με ενίο τουλάχιστον τρόπο, με εναρμονισμένο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους σε σχέση με το συντονισμό της διαδικασίας και την πρόθεση των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων στα κράτη-μέλη. Επίσης, υπογραμμίζουμε στη γνωμοδότησή μας εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης το σημαντικό ρόλο της πολιτικής συνοχής σε αυτή τη διαδικασία ανάκαψης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι η κατεξοχήν αναπτυξιακή πολιτική για την Ένωση αυτή η πολιτική, η πολιτική συνοχή. Θα πρέπει να εμβαθυνθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμεινού ώστε να έχουμε ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επενδύσεων για την ε, πολιτική συνοχή και μεγαλύτερα ε, ποσοστά επενδύσεων. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο τονίζουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει πιο γρήγορη εφαρμογή ε, των έργων στο πλαίσιο του ΕΦΣΥ. Γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν συντονιστικές δομές για να αξιοποιήσουν σωστά τα κονδύλια της συνοχής. Επίσης, ό,τι αφορά αυτό το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, να επικοινικύνθηκε ως προς την διάρκεια ισχύω του και έτσι θα προωθηθούν περισσότερες επενδύσεις και θα αναπτυχθούν συνέργειες και συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων ταμείων και εργαλείων. Αυτό θα οδηγεί σε βελτίωση. Και τονίζουμε το ρόλο του προγράμματος για την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν ε, λοιπόν βοήθεια για να φέρουν σε πέρα σε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις. Τονίζουμε ότι είναι σημαντικό να είναι βιώσιμες αυτές οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο και θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τις επιχειρήσεις, για τις επενδύσεις πρέπει να βελτιωθούν ε, οι προϋποθέσεις και το πλαίσιο. Αυτά είναι συντομία σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας και τώρα βέβαια περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω την άποψη των ασκιωδών εισηγητών γιατί βέβαια μαζί θα καταρτήσουμε μια καλή γνωμοδότηση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στους σκιώδες ζητές και συγκεκριμένα καταρχάς τον κύριο Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εν συντομία, σε σχέση με τη γνωμοδότησή σας, θα ήθελα να τοποθετηθώ και να πω ότι πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι Έχετε περιγράψει ουσιαστικά συντομία όλες τις προτεραιότητες που άπτονται του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα καταθέσω σχετικά κάποιες τροπολογίες για μικρές αλλαγές. Θα μιλήσω για την ανεργία κυρίως και για το ρόλο του Ταμείου ΕΦΣΥ, Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά το ΕΦΣΥ συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποια ανισορροπία. Το είχαμε αναφέρει και στην τελευταία μας έκθεση. Ανισορροπία λοιπόν μεταξύ των 15 ε, και 13 χωρών μελών της Ένωσης. 91 προς 9% ήταν ο λόγος. Δηλαδή ωφελούνται πολύ περισσότερο τα παλαιότερα κράτη ενώ Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει φέτος και ποια είναι η αναλογία μεταξύ ε, των δύο αυτών ομάδων χωρών. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια σημαντική παρατήρηση που θα πρέπει να ληφθεί. Υπόψη και η δεύτερη παρατήρηση μου αφορά την ανεργία. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ε, αναφέρεστε στα ποσοστά ανεργίας των νέων είναι βαθιές οι ρίζες της ε, ανεργίας και σίγουρα η ε, πολιτική συνοχή ε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταπολέμηση του φαινομένου της ανεργίας. Πιστεύω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της δομικής ανεργίας και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτά είναι τα δύο βασικά ζητήματα για τα οποία θα ήθελα να επιφέρω ε, κάποιες βελτιώσεις, κάποιες ε, τροπολογίες για να συμπληρώσω αυτά που αναφέρετε εσείς. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πυρίνης και είναι ο επόμενος. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι η έκθεση για την, μάλλον η επισκόπηση για την ανάπτυξη και νομοδότης της δικής μας ε, Επιτροπής θα πρέπει να δοθούν σε σχέση και με την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Και πρέπει να πω ότι και οι τρεις αυτές εκθέσεις ε, προσλαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερη βαρύτητα. Τις ε, τελευταίες ημέρες βλέπουμε να υπάρχουν ανησυχητικές Ε, δηλώσεις και ε, εξέλιξεις σε σχέση με την οικονομία. Οι πολιτικοί ηγέτες εχθές ε, εξέφρασαν ανησυχίες και στον Ταβός σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και πραγματικά οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές θα εμβαθυνθούν λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προβούμε σε, έναν εκβάθρονα, σε μια εκβάθρονα αναθεώρηση των πολιτικών μας. Η γνωμοδότησή σας πάντως αποτελεί μια καλή βάση εργασίας για την ε, περαιτέρω διατύπωση προτάσεων για να έχουμε πραγματικά ποιοτικέ αλλαγές που θα έχουν νόημα, που θα έχουν σημασία. Το policy mix είναι σημαντικό. Τι πολιτικές θα εφαρμόσουμε. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό μείγμα πολιτικών για να μπορέσουμε να λάβουμε τις σωστές πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις για να υπάρξει βελτίωση των δικτών της ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα. Αυτά δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε. Οπότε χρειάζονται ακόμα περισσότερα μέτρα, γιατί αυτές οι βελτιώσεις δεν αρκούν. Και αυτή η εμβάθυνση. Έχουμε ένα τρίγωνο του διαβόλου, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι. Χρειάζονται νέες αρχές, νέες ε, κατευθυντήριες γραμμές. Έχουμε τον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος επίσης ε, προσλαμβάνει και μεγαλύτερη σημασία. Η επενδυτική πολιτική επίσης θα πρέπει ε, να αναθεωρηθεί εκ βάθρων. Στην εκθέση της Επιτροπής ΕΚΟΝ Γίνεται λόγος και για τις δημόσιες επενδύσεις που σημειώνουν πτώση. Και δυσκολεύει η κατάσταση ε, στις περιφέρειες. Υπάρχουν ομάδες ε, που είναι κοινωνικά αποκλεισμένες. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση της δικής μας Επιτροπής θα μπορούσε να πει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό το θέμα. Αναφέρατε το πρόγραμμα στήριξη των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων που αναμφίβολα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όμως το πρόγραμμα αυτό να εστιάσει στις προτεραιότητες ε, του, που έχουν να κάνουν με την καλύτερη χρήση του ΕΦΣΙ και των διαθροτικών ταμείων. Οι ταστικέ μεταρρυθμίσεις μπορούν να εμπνευθούν ποικίλο τρόπο όπως γνωρίζουμε όλοι. Ουσιαστικά πρέπει να αντιμετωπιστούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται και με τη μη καλή απορρόφηση των κονδυλίων. Πιστεύω ότι για να έχουμε καλές επενδύσεις χρειάζεται να ξανασκεφτούμε και την επενδυτική πολιτική, να την επικαιροποιήσουμε. Επίσης έχουμε μιλήσει για την ποσοτική χαλάρωση και μιλήσαμε για διάφορες αλλαγές. Τώρα πιστεύω πρέπει να στραφούμε στην ποιότητα πέραν της ποσότητας για να έχει απήχηση όλα αυτή και στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σομαριζέ. Κύρια Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δώσατε έμφαση στο θέμα της ενεργείας των νέων που παραμένει εξαιρετικά σημαντική σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης, ιδιαίτερα στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές και παρά την οικονομική ανάκαμψη, την ισχνή στην Ευρώπη, αυτή η τάση δεν φαίνεται να αντιστρέφεται στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Εμένα μου αρέσει να συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την περιφερειακή πολιτική, εδώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εμείς πάντα θεωρούσαμε ότι αυτό δεν έχει σχέση με την περιφερειακή πολιτική. Αυτές οι συστάσεις αναχώρα και οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, ουσιαστικά νοθεύουν την περιφερειακή πολιτική. Είμαστε άλλωστε πεπισμένοι ότι αυτές οι διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτές οι πολιτικές λιτότητας, είναι αυτές που συνεισέφεραν τα μάλα για να επιδεινωθεί η οικονομική και η κοινωνική κατάσταση στο σύνολο της Ευρώπης και δεν πρέπει να αναπαράγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Υπάρχει δηλαδή μια σημαντική απόκληση εδώ μεταξύ μας. Κατά τα λοιπά βεβαίως συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τον κύριο Σκάρλετς, ε, ο κύριος Ρόπε θα μιλήσει στο όνομα της ομάδας του. Ευχαριστώ Πρόεδρε να πω και εγώ δύο λόγια. Οι προτάσεις σας ε, αφορούν κάποιες, κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα. Ε, βεβαίως τη στιγμή υπάρχει μια οικονομική ανάκαμψη, όχι επαρκής, όχι με επαρκείς ρυθμούς, αλλά οι επιπτώσεις της κρίσης του 2008 δεν έχουν ε, αντισταθμιστεί από τους ρυθμούς ανάπτυξης. Σε πολλές χώρες ε, οι πολίτες ακόμα ζουν τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής, ε, έχουν χαμηλά εισοδήματα, υπάρχουν κάποιες θετικές τάσεις. Θα ήθελα να πω ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεισφέρει περισσότερο στην ανάπτυξη των τοπικών περιφερειακών οικονομιών. Η πολιτική συνοχής συχνά ε, έχει ως σκοπό ε, τη δημιουργία δημοσίων αγαθών, τη βελτίωση των δημόσιων υποδομών, αλλά πρέπει να έχουμε και καλύτερα εργαλεία ε, στη διάθεση των περιφερειών. Πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες της περιφερειακής πολιτικής με πιο ευέλικτο τρόπο. Οι τοπικές αρχές θα πρέπει να μπορούν και αυτές να συνεισφέρουν σε καλά project και αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης σε μια σειρά από περιφέρειες. Στο μέλλον η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ειδωθεί ε, ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο υποστήριξης τοπικών πρωτοβουλειών που θα επιτρέπει ένα ε, κάποιο επίπεδο ευελιξίας. Τώρα υπάρχει το θέμα της ενέργειας γνωρίζουμε ότι τα κράτη-μέλη αγοράζουν τη μισή τους περίπου ενέργεια από τρίτες χώρες. Μιλάμε για 400 δισεκατομμύρια το χρόνο αξία. Θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε οι ίδιοι να παράγουμε ενέργεια, να χρησιμοποιήσουμε τοπικούς πόρους γι' αυτό. αγοράζοντας ενέργεια αλλού συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη, στους ρυθμούς ανάπτυξης τρίτων χωρών ε, και αυτές οι χώρες ε, δεν χρησιμοποιούν αυτή την ανάπτυξη, αυτά τα κέρδη ε, με φιλικό τρόπο προς την Ευρώπη. Είναι περίπλοκα τα πράγματα. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας την κυκλική οικονομία, ένα χρήσιμο εργαλείο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των πλέον μειονεκτούσων περιοχών. Συχνά διαπιστώνουμε ότι ε, οι μεγαλύτερες πόλεις ε, έχουν ένα πλεονέκτημα ε, και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Στη χώρα μου, στη Λιθουανία, η διαφορά επίπεδου ζωής ε, είναι τη τάξη του 1 προς 3 ανάμεσα στην πρωτεύουσα και την Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να πιέσουμε, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε αυτό το χάσμα. Σημαντικό και αυτό το στοιχείο. Ε, θα συμβάλλει γενικότερα στην προσπάθεια σύγκλησης που γίνεται. και δεν θα έχουν την ε, τάση ή τον πειρασμό, αν θέλετε, οι πολίτες ε, κάποιων χωρών να μεταναστεύουν σε άλλες. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα των φορολογικών συστημάτων σε κάποια κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ισότητα. Υπάρχουν πολλά ασύμβατα στοιχεία σε ό,τι αφορά φορολογικό σύστημα κάποια κρατημέλη ε, προσπαθούν να προσελκύσουν ε, μέσα στο φορολογικό του συστήματος ε, μια σειρά από εταιρείε και άλλες χώρες ε, ζημιώνονται από αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε δεν πρέπει να ξεχνάμε το φορολογικό ζήτημα πρέπει και αυτό να είναι μέρος της ατζέντα μας ευχαριστώ πολύ δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλο το λόγο από τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζιο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον εκπρόσωπο, στην εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή επιτροπή. την κυρία Λάκοβα. Είναι εδώ κυρία Λάκοβα. Βεβαίως, παρακαλώ. Uh, yes, I would uh, like to thank you for... Σας ευχαριστώ για την γνωμοδότηση. Για τα ωφέλη που προκύπτουν από τα κονδύλια. Πιστεύουμε ότι σωστά επιδιώκει την κατάλληλη κατεύθυνση η έκθεση αυτή. Έχουμε κάποια σχόλια για το γεγονός ότι οι συστάσεις ε, αλλοιώνουν την πολιτική. Αυτό θέλουμε να το σχολιάσουμε. Δεν ισχύει, πιστεύουμε, ότι οι συστάσεις αναχώρα αλλοιώνουν την πολιτική. τα κάτι μέλη πρέπει να κάνουν προσπάθειες για να εκτελούνται καλύτερα τα διάφορα κονδύλια, να χρησιμοποιούνται καλύτερα τα κονδύλια. Ε, τα διευθυντικά ταμεία ε, πρέπει να, να διαθέτουν ε, με τον σωστό τρόπο βάσει των συστάσεων αναχώρα τα κονδύλια στην κάθε χώρα. Όμω οι συστάσει πολλέ φορέ έχουν πολύ μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οπότε οι χώρε γνωρίζουν πολύ καλά τι ε, κονδύλια θα λάβουν και τι όφελο πρέπει να παραχθεί για του πολίτε. Τα διαδοτικά ταμεία επίση έχουν πολύ σωστά συνδυαστεί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τη συνοχή, όχι μόνο με, την, ε, με τις που γίνονται, αλλά και με την ερεσιμότητα εξάντε που έχει μελετηθεί ένα χώρα. Και έτσι μόνο αν εκπληρώνονται μόνο αυτή η ρεσιμότητα και μόνο αν ε, έχει ε, προλεμβεί το έδαφος για να αξιοποιηθούν οι επενδύσεις θα μπορέσουν τα προγράμματα δράσης να εφαρμοστούν σωστά. Εάν το επενδυτικό το οποίο στα κάτι μέλη που έτοιμαστε σωστά θα γίνει και ε, έφορο για να μπορέσουν οι επενδύσεις αυτές να φέρουν άντηση και να υπάρξουν βιώσιμα αποτελέσματα και να μην υπάρξει μαρασμός μετά το τέλος των επενδύσεων. Νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, όμως ε, οι συστάσεις δεν αλλοιώνουν την πολιτική. Ε, ίσα ίσα μπορούν να συνδυαστούν και να καλύψουν ανάγκες στα κράτη-μέλη, καθώς και να αξιοποιηθούν στο κατάλληλο πεδίο για να αξιοποιηθούν σωστά και επενδύσεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Σομαρζέ θέλει να κάνει μια σύντομη παρατήρηση. Ναι, μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Παρακολουθώ αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σημειώνω, αλλά εδώ είμαστε πολιτικό σώμα και είμαστε και μια κοινοβουλευτική επιτροπή όπου διεξάγονται πολιτικές συζητήσεις. Έχουμε λοιπόν το δικαίωμα να αποτιμήσουμε όπως θέλουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και αυτή τη στιγμή λέω ότι οι συστάσεις αυτές αναχώρα και ο σχεδιασμός, η ένταξη της ε, περιφερειακής πολιτικής ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλοιώνουν το χάραξη πολιτικής, αυτό είναι πολιτική θέση. Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου ε, αντιπαρατάσει τη δική της θέση ως προς αυτό, προφανώς είναι η άποψή μου. Ευχαριστώ ως εισηγήτρια και της έκθεσης αυτής και πρόεδρος της Επιτροπής ε, δεν μπορώ παρά να σεβαστώ τις πολιτικές απόψεις όλων των πολιτικών ομάδων οι οποίες έχουν βεβαίως την ε, θέση που τους αρμόζει και θα απηχηθεί αυτή στην ε, τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ρέτζη. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους και εισηγητές για τις συνεισφορές τους και τώρα θα περιμένω τις προτάσεις σας για τροπολογίες. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, από την Γενική Διεύθυνση Ρέντζιο ε, για την τοποθέτησή της. Γνωρίζουμε την ε, θέση αυτή γενικώ. Καταγράφουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις, θα τις λάβουμε υπόψη, όμως η τελική γνωμοδότηση της Ρέτζη θα είναι βεβαίως αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών όλων των εισηγητών και σκιωδών εισηγητών. Σας ευχαριστώ πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι στις 30 Ιανουαρίου την επόμενη εβδομάδα, όπως προείπα. Ευχαριστώ. Να προχωρήσουμε τώρα. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη σεμινάριο που οργανώθηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής B για την 7η έκθεση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Το εργαστήριο αυτό το είχε οργανώσει η υπηρεσία του τμήματος Β κατόπιν ετήματος της Επιτροπής μας για να προσφέρει την συμβολή του την σύνταξη της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής επί της έκθεσης ε, συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 7η ε, παριθμών που υιοθετήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Όπω βλέπετε και στο πρόγραμμα, ε, το πάνελ των εμπειρογνωμόνων συμπεριλαμβάνει προσώπου των πανεπιστημίων αλλά και άνθρωπους που στην πράξη ασχολούνται με θέματα αυτά από το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα ασχοληθούμε με την μελλοντική εξέλιξη του τι συμβαίνει σε εδαφικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με βασικά ζητήματα όπως η πάγιδα του μέσου εισοδήματο, η αστική διάσταση της Επιτροπής Συνοχής, η ατζέντα για τα αστικά κέντρα, οι σχέσεις μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών τη υπαίθρου, η εξισορρόπηση ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων και εδαφικών αναγκών. Εδώ υπάρχει μια σειρά από έγγραφα που έχουν ε, αποσταλεί τους ε, βουλευτές της Επιτροπής ΡΕΤΖΙ. Εάν δεν τα έχετε, μπορείτε να τα βρείτε κάπου στην αίθουσα. Α, στο βάθος, όντως. Και έχετε και το πρόγραμμα, λογικά, του εργαστηρίου. Να ξεκινήσουμε να κηρύξω την έναρξη του εργαστηρίου δίνοντας το λόγο στον κύριο Ζουλό, ο οποίος είναι εισηγητής για την 7η έκθεση με θέμα την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ρέντζη ε, η οποία είναι ιδιες πρωτοβουλιας της επιτροπης ρεντζη έκθεση για τη δική μας ε, την Επιτροπή. Οπότε το λόγο έχει ο κύριος Ζουλό. Euh. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εισαγωγικά κάποιε παρατηρήσει πριν ξεκινήσει το εργαστήριο. Θέλω να ευχαριστήσω εκ των προτέρων του προσκεκλημένου μα που απεδέχθησαν την πρόσκληση και θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια. Όπω είπατε, είμαι ο συντάκτη ε, τη έκθεση για την 7η έκθεση συνοχή. Γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα ότι είναι πολύ ε, στενό τον επόμενο μήνα θα παρουσιάσω την έκθεση μου στην Επιτροπή μας και ο στόχος μου είναι να στείλω ένα σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν κατατεθούν οι προτάσεις ε, για το προσεχές πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν θέλω να είναι ένα άχρωμο άοσμο σχέδιο έκθεσης ε, και πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντλήσουμε διδάγματα από την πολιτική συνοχής για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα και προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής στο μέλλον. Φαντάζομαι ότι θα αναλύσουν οι εμπειρογνώμονες ε, ε, τα θέματα που έχουν αναλάβει να μας παρουσιάσουν και τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, όπως για παράδειγμα η παγίδα του μεσοδήματος όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν. εντοπίζονται το πρόβλημα, τώρα πρέπει να βρούμε λύσεις. Εγώ αποδίδω σημασία στο θέμα και θα με απασχολήσει και στην έκθεσή μου. Το δεύτερο είναι οι αστικές προκλήσεις. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Οι πόλεις ε, παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Υπάρχουν θύλακες φτώχειας σε ορισμένε από αυτέ τι πόλεις. Ενώ δίπλα έχουμε άλλες περιοχές ε, που δείχνουν ε, επιτυχία. Επίσης, οι προτεραιότητες, οι στρατηγικές ε, δεν θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την εδαφική διάσταση που είναι επίσης σημαντική. Και βέβαια έχουμε και την απλούστευση. Πολλά έχουμε πει για την απλούστευση. και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την άποψη των ερετών ε, επιτόπου για να διαμορφώσουμε την άποψή μας για το μέλλον. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα πραγματευτώ στην έκθεσή μου. Το καλύτερο όμως νομίζω είναι να ακούσουμε ευθύ αμέσω ε, τους ομιλητές μας για τα κρίσιμα αυτά θέματα που από της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Επομένως, αρχίζει η συζήτηση και έχω την ε, χαρά να δώσω το λόγο στον καθηγητή Αντρές Ροντρίγκεθ Πόσε, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας ε, στο Τμήμα Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος από το London School of Economics. Θα μας παρουσιάσει το θέμα περιφερειακή παγίδα μεσισοδήματο και η πρόκληση για τον οικονομικό δυναμισμό της Ευρώπης. Ε, κύριε Ροντρίγκεθ, πώς έχετε το λόγο. 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα και βεβαίω να συζητήσουμε και το σημαντικό κείμενο του 7ου, της 7 Υπάρχουν, ε, Υπάρχουν δύο τύπου περιφέρειες που έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτικών ηθινών και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Αφενό, έχουμε στι λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ που έχουν το χαμηλότερο επίπεδο ε, κατά κεφαλήνα ΑΕΠ και έχουμε από την άλλη τις μεγάλες μητροπόλεις, τα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης. Ε, βεβαίως πρόκειται για δύο πολύ σημαντικά μέρη της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης της Ένωσης. Όμως υπάρχουν και άλλοι τύποι περιφερειών, τις οποίες έχουμε κάπως παραμελήσει. Αυτές που βρίσκονται κάπου στη μέση, σε αυτό το, τη μέση, την παγίδα μέσου εισοδήματο. Πρέπει να δείξουν και αυτές ότι έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Για ποιες περιφέρειες μιλάμε. Χαρακτηρίζονται ε, βεβαίως ε, όχι από ομοιογενή χαρακτηριστικά, ε, Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία μοιράζονται. Αφενός, εάν δείτε αυτό το χάρτη, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για περιοχές που τα τελευταία 25 χρόνια είχαν ε, σταθερά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση ε, με τις ε, μεγάλες μετροπόλεις αλλά και τις μειονεκτούσες περιοχές. Είναι για, μιλάμε για περιφέρειες που φτάσαν σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης λίγο πιο κάτω από το μέσο όρο της Ένωσης και έχουν μείνει εκεί, στάσιμες, ή που στο παρελθόν ήταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έκτοτε έχουν μια σταθερή μείωση. Αυτό αποτυπώνεται και σε άλλες μορφές οικονομικής ανάπτυξης, ε, χαμηλή ρυθμή απασχόλησης. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε στη Νότια Ιταλία, στη Βορειοανατολική Γαλλία, στη Βαλονία, στο Βέλγιο. Είναι περιοχές που δυσκολεύτηκαν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης ε, για τον τοπικό τους πληθυσμό. Και επιπλέον ε, στις περιφέρειες αυτές ε, είχαμε χαμηλή απόδοση ε, σε ό,τι αφορά την το υπόλοιπο της χώρας. Δηλαδή ε, είναι έχουν χαμηλά επίπεδα απόδοση. Ε, ανέκαθεν και πριν την κρίση. Εδώ βλέπετε την απόδοση σε σχέση με το μέσο όρο της κάθε χώρας ε, τα τελευταία 25 χρόνια. Ε, επίσης ε, ε, υπάρχουν χώρες που έχουν θεσμικά προβλήματα διακυβέρνησης, διαφθοράς, αποτελεσματικότητας της, ε, των κρατικών αρχών. Ε, δείκτες που είναι χαμηλότεροι σε σχέση με αυτό που θα ανέμενε κανείς. Πώς έχει προκύψει λοιπόν αυτή η παγίδα του μέσου εισοδήματο. Ε, στο παρελθόν ε, έχουμε, μιλάμε για χώρες που είχαν αρκετά γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης, φτάσανε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο βιωτικό και μετά κόλλησαν εκεί. Γιατί? Ε, διότι είχαμε μια αύξηση των εισοδημάτων στο παρελθόν και αυτές οι χώρες έγιναν ακριβές. Έγιναν ακριβές για να μπορούν να ανταγωνιστούν ε, στην κλίμακά τους ε, σε επίπεδο παραγωγής σε σχέση με άλλες πιο ελκυστικές περιοχές ακόμα και είναι λιγότερο ανεπτυγμένες αλλά και με άλλες περιφέρειες ανά τον κόσμο που μπορούν να προσφέρουν τα, τα ίδια προϊόντα με την ίδια ποιότητα σε πολύ χαμηλότερο κόστος. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι πολλές από τις περιφέρειες αυτές δεν είναι σε ένα επίπεδο που να μπορούν να παρέχουν ε, τα πλεονεκτήματα που παρέχουν οι μεγάλες μητροπόλεις ε, σε επίπεδο σύνδεσης, ε, σε επίπεδο επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και περιβάλλοντων και σε επίπεδο της δυνατότητας καινοτομίας και χρησιμοποίηση των δεξιοτήτων που βρίσκονται εκεί. Αυτές οι περιοχές λοιπόν είναι ε, έτσι κάπου στη μέση. Είναι στριμωγμένες. Δεν μπορούν να αντικανονιστούν σε επίπεδο κόστους διότι βρίσκονται, είναι, πολύ, είναι υπερβολικά κεντρικές αλλά δεν είναι αρκετά κεντρικές για να είναι ανταγωνιστικές. Αυτές οι περιφέρειες λοιπόν αρχίζουν να βιώνουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες. Και αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση. Αφενός οι περιφέρειες αυτές έχουν δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης, δυνατότητες που δεν χρησιμοποιούνται, που δεν, που εκμεταλλευόμαστε και επίσης ε, αυτή η δυσαρέσκεια εκφράζεται. Ε, εκφράζεται εκλογικά σε πολλές χώρες. Στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, ίσως και περισσότερα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, το έχουμε διαπιστώσει και στις ΗΠΑ αλλά και αλλού στον κόσμο, στην Ταϊλάνδη ε, μεταξύ άλλων. Γιατί αυτή η γεωγραφία της δυσαρέσκειας ε, εμφανίστηκε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Στις περιφέρειες αυτές δεν έχουμε κάτι κάτι για αυτές. Δεν είναι ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ε, έχουν λάβει χώρα σημαντικές επενδύσεις. αλλά οι επενδύσεις αυτές, με κάποιες εξαιρέσεις, δεν ήταν αποτελεσματικές. Σε εθνικό επίπεδο είχαμε μεταφορά ε, και ενίσχυση από το κράτος πρόνοιας, αλλά αυτό οδηγεί σε μία εξάρτηση από τις... μια ε, ε, εξάρτηση μάλλον, σε μια, ένα καθώς εξάρτηση για αυτές τις μια εξαρτηση μαλλον σε μια ενα εξαρτηση για αυτες τις περιφερειες δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης ε, δημόσιες, ε, ε, έχουν συνήθως υψότερα ποσοστά δημοσίων θέσεων εργασίας σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις αλλά και σε σχέση με τις πιο μειονεκτούσες περιοχές αλλά αυτό δεν αρκεί για να μπορέσει να πυροδοτήσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, μη χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων. Πολλές πολιτικές στο παρελθόν δεν ήταν ε, αποτελεσματικές, ορισμένες φορές ήταν λανθασμένες, ε, ε, βασίστηκαν στις παλιέ βιομηχανικές δομές ε, που δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν δίκτυα που να παράγουν μια αλλαγή αξίας. γενικά υπήρξε μια κακή διαχείριση. Αυτή τη στιγμή οι περισσότερε από τι πολιτικές έχουν συνεισφέρει είτε στην διατήρηση του παρόντος επίπεδου εισοδημάτων. Ε, καλές είναι οι κοινωνικές πολιτικές, αλλά από μόνες τους δεν αρκούν. Εδώ μιλάμε για απλά για κοινωνικές πολιτικές χωρίς μια στρατηγική. Και αυτό δείχνει ότι σε πολλέ από τις περιφέρειες δεν υπάρχει πραγματικό μέλλον. Ε, δεν υπάρχουν δυνατότητες, δεν υπάρχει δυνατότητα κάποιο να βρει μια θέση εργασία που να το επιτρέψει να ευημερήσει μακροπρόθεσμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, είναι ε, ορατό και είναι απτό ε, μαζικά στους πληθυσμού των περιοχών αυτών. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε προ μια διαφορετικού τύπου πολιτικής. Πολιτικές ε, που να φέρουν πιο ψηλά στην ατζέντα αυτέ τι περιοχέ με την παγίδα του μέσου εισοδήματο. Γιατί, γιατί υπάρχει σημαντική οικονομική ανάγκη. Πολλές από τις περιφέρειες αυτές εκπροσωπούν ένα σημαντικό ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να του δοθούν περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που έχουν τώρα. Επίσης οι περιφέρειες αυτές έχουν σημαντικές οικονομικέ δυνατότητε σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ε, ακαδημαϊκές αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΩΣΑ έχει προκύψει ότι ναι βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1 τρίτο της ανάπτυξης προέρχεται από τις, τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα 2 τρίτα όμως έρχονται από αλλού και ένα μεγάλο ποσοστό αυτού προέρχεται από αυτά, αυτές τις περιφέρειες μέσου εισοδήματος που είναι έχουν μπει σε αυτή την παγίδα. Είναι, πρόκειται και περιφέρειες που στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ε, σημαντική ανάπτυξη για την Ευρώπη. Και δεν μπορεί η Ευρώπη ε, να παραμελήσει αυτές τις δυνατότητες ανάπτυξης. Από την άλλη πρέπει να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε την ε, ε, ανάπτυξη αλλού στην Ευρώπη. Είναι ένα σύστημα ε, αλληλεξαρτήσεων. Ε, η ανάπτυξη στις, ε, μεγάλες, στα μεγάλα αστικά κέντρα εξαρτάται από την ανάπτυξη στις περιοχές μέσου εισοδήματο. Δηλαδή το να παραμελήσουμε ένα μέρος του συστήματος, να το αφήσουμε στην άκρη, διακυβεύει το σύνολο του συστήματος. Το έχουμε δει αυτό στην Ευρώπη οι δυνατότητε ε, των μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των λιγότερων των πιο περιοχών ε, μειώνονται εφόσον παραμελούμε τις υπόλοιπε. Δεν είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πολιτικές, χρειαζόμαστε καλύτερες πολιτικές ε, και διαφορετικές. Πολιτικές που απομακρύνονται από μια απλή ατζέντα κράτου πρόνοια, α πούμε ε, και κοινωνικής ε, στήριξης που δεν θα βοηθήσουν μακροπρόθεσμα να απομακρυνθούμε από τα απλά, απλά να προστατεύουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, και να μην τους δίνουμε τη δυνατότητα ουσιαστικά να ανταγωνιστούν και να ε, πρωταγωνιστήσουν στις νέες, οικονομ... στις νέες μορφές Χρειαζόμαστε πολιτικές ε, που θα δημιουργούν διοξιότητες, θα δημιουργούν δυνατότητες, θα δημιουργούν ένα περιβάλλον, ένα οικοσύστημα ε, που να είναι ευνοϊκό για την καινοτομία και για την παραγωγικότητα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Υπάρχει μια ιδέα, μια θεωρία αν θέλετε, σύμφωνα με την οποία χρειαζόμαστε πολιτική, πολιτικές που να μην είναι ενιαίες ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που ε, να ε, λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του καθένα. Πολιτικές δηλαδή που να μην βασίζονται σε κάποιες γενικές αρχές που θα εφαρμόζουμε ομοιογενώς αλλά που θα βασίζονται σε στοιχεία σε δεδομένα που θα βοηθούν στην προσαρμογή στα χαρακτηριστικά ε, της κάθε περιφέρειας και ιδιαίτερα των αυτών των περιφερειών ε, μέσω εισοδήματο. Ο στόχος πάνω απ' όλα είναι να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις τοπικές δυνατότητες που παραμένουν αχρησιμοποιητές. Πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι κανείς ε, δεν πρόκειται να μείνει πίσω. Κανείς δεν θα πρέπει να ε, νιώθει ότι μειονεκτεί ανάλογα με το που έχει γεννηθεί. Πρέπει οι δεξιότητες να μπορούν να μεταφερθούν. Αυτή τη στιγμή πολλοί κατοίκοι, κάτοικοι αυτών των περιοχών ε, είναι κάπως παγιδευμένοι εκεί. Δεν μπορούν, δεν έχουν δεξιότητες να ε, να προχωρήσουν. Πρέπει οι ίδιοι να έχουν τη δυνατότητα και να κάνουν την επιλογή αν θα μείνουν στην περιοχή τους, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξή της ή ε, εάν με τις δεξιότητες που θα μπορέσουν ε, να αποκτήσουν θα πάνε αλλού. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε βεβαίως την αναποτελεσματικότητα, τα σημεία συμφόρησης που περιορίζουν την ανάπτυξη ε, και τι δυνατότητε ανάπτυξη πολλών, πολλών εκ των περιοχών αυτών. Δεν έχω το χρόνο να μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε, εάν πάντως ε, ενδιαφέρεστε υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που μπαίνουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε. Λέω μπαίνουμε διότι συμμετέχω μαζί με άλλου στην σύνταξη του κειμένου αυτού για το πώ μπορούμε να πετύχουμε αυτού του στόχου. Θα ήθελα τέλο να πω ότι αυτή τη στιγμή ξεχνώντας αυτές τις περιφέρειες μέσω εισοδήματο, η Ευρώπη δημιουργεί προβλήματα στον εαυτό της. Πολλές δυνατότητες ανάπτυξης αυτή τη στιγμή υποχρησιμοποιούνται. Και αυτό, αυτές οι δυνατότητες μεταφέρονται αλλού στον κόσμο. Δεύτερον, αυτές οι περιφέρειες έχουν σημαντικές δυνατότητες να επηρεάσουν την εφημερία και άλλων περιοχών και τρίτον, αυτή η αίσθηση ε, ανησυχίας και δυσαρέσκειας ε, τα οικονομικά προβλήματα θα δημιουργήσει μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα αλλά και κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Κάτι που θα υπονομεύσει όχι μόνο την ευημερία αυτών των περιφερειών αλλά και την ευημερία και τις δυνατότητες ανάπτυξης της Ευρώπης στο σύνολό τη. Δεν μπορεί, δεν έχει το δικαίωμα η Ευρώπη να παραμιλήσει αυτές τις περιφέρειες θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις περιοχές ε, που βρίσκονται στην παγίδα του μέσου εισοδήματος. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. I'm sure there... Ευχαριστούμε. Είμαι βεβαία ότι θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις στη συζήτησή μας μετά, αλλά τώρα να, συνεχίσουμε με την επόμενη παρουσίαση. Πώς να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των αστικών κέντρων. Δυναμικές τάσεις, τοποθετήσεις και διαμόρφωση της πολιτικής συνοχής μας. Ο ομιλητής μας θα είναι ο Μαρτ Γκρίζελ, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου ε, Αστικής Γνώσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον σεμινάριο να ξεκινήσω παρουσιάζοντας το δίκτυό μας σε όσους δεν το γνωρίζουν. Είμαστε ένα δίκτυο κρατών μελών που συνεργάζονται από κοινό για διάφορα ζητήματα ώστε να υπάρχει μια διεπαφή μεταξύ των ερευνητών, των όσων χαράζουν πολιτική και των όσων εργάζονται με τα θέματα αυτά στην πράξη. Οι μελέτες μας είναι λόγω χάρη αυτοί που δημοσιεύσαμε πέρσι για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων σε 35 χώρες στην Ευρώπη και εκτός. Οργανώνουμε διασκέψεις με συμμετοχή των μελών μας για την παγκοσμιοποίηση λόγου χάρη, για την εξισορρόπηση των αναγκών αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης σε διάφορες χώρες. Ε, είδαμε επίσης το σύμφωνο του Άμστερνταμ και την προσαρμογή του μετά από την παρέμβαση της Ολλανδικής Προεδρίας το 2016. Έχουμε... Πάω πίσω στη διαφάνεια Έχουμε διοργανώσει πολλά σεμινάρια και συνεδριάσεις, διασκέψεις, ημερίδες ανάλογα με τις εταιρικέ σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ατζέντα για την καταπολέμηση της φτώχειας, την υποδοχή των προσφύγων, προσφύγων και μεταναστών, τη χρήση της γης, θα θυμίσω στους Ισπανούς συναδέλφους επίσης την Ισπανική αστική ατζέντα ή την περιφερειακή πολιτική και την εφαρμογή της στην Κύπρο καθώς και την κοινωνική ένταξη που αναπτύξαμε με συναδέλφους από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να μιλήσω για την διάσταση των αστικών κέντρων στην πολιτική συνοχή. Δεν είναι κάτι το καινούργιο. Είναι μια καινούργια τάση ε, που έχει δυναμικό χαρακτήρα και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνέ επίπεδο. Και ήδη μας έχει απασχολήσει. Ήδη από το 2016 ξεκίνησε να έχει μεγάλη ε, απήχηση με την ε, έγκριση της ατζέντα ε, την άνοιξη του 2016 με την επίδραση της Ολλανδικής Προεδρίας και το φθινόπωρο του 2016 με την έγκριση των βιώσιμων στόχων. Υπάρχουν πολλά σχετικά εργαλεία που προβλέφθηκαν στο πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 τα γνωρίζετε και δεν θέλω να αναπτύξω αυτά σήμερα. Αυτό που θέλω είναι να σας παρουσιάσω την αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Εδώ έχω δύο παραμέτρους να αναπτύξω. Ως διευθυντής του δικτύου αλλά και ω ε, άνθρωπο που ασχολούμαι πάρα πολύ με τα αστικά κέντρα και τι εταιρικέ σχέσει που απαιτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να παρουσιάσω έναν τρόπο συνεργασία επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συμμετέχουν πολλοί εταίροι και πολλοί ενδιαφερόμενοι, πολλά αστικά κέντρα και μπορούμε να βασιστούμε στα εργαλεία και τις εμπειρίες από συγκεκριμένα αστικά κέντρα. Η αστική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το σύμφωνο του Άμστερνταμ, ε, εάν μελετήσετε τα κείμενα, θα σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες για το όλο ζήτημα. Μιλάμε για ζητήματα πολυθεματικά, τα οποία όλα μπορούν να αξιοποιηθούν και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να επικεντρωθούμε στα θέματα προτεραιότητας που αναφέρει και το σύμφωνο του Άμστερνταμ. Οι πρώτες εταιρικές σχέσεις 4 ως 6 που έχουν εφαρμόσει τα προγράμματα δράσης τους είναι αυτές τις οποίες θέλω να σταθώ. Ασχολούνται με την καλύτερη νομοθεσία, την καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και την καλύτερη χρηματοδότηση. Και μπορούν να δώσουν σημαντική συνεισφορά για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Θα θίξω μερικά από τα κύρια ζητήματα όπως η ευελιξία, η απλούστευση και η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής οι ουσιαστικέ διασυνδέσεις. Δεδομένου του περίπλοκου του θέματος, απλώς θα σκεγγραφίσω τις αδρές γράμμες της πρότασης. Δεν έχουμε χρόνο για κάτι περισσότερο σε αυτό το εργαστήριο. Με τις προτάσεις που έγιναν για μεταρρύθμιση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν εκφράστηκε παρόλα αυτά η επίσημη θέση του δικτύου μας ή άλλων. Αυτό που μας, που μας απασχόλησε να μελετήσουμε είναι η μακροοικονομική αιρεσιμότητα ή τα διάφορα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την πολιτική συνοχή σε σχέση με την αστική διάσταση και τι είναι διαθέσιμο από τα κρατικά κονδύλια, το κρατικό κορβανά στα διάφορα κρατημέλη. Αυτό που δεν θα σα ευνηδιάσει είναι ότι όλες οι μέχρι τώρα εξελίξεις τονίζουν τη σημασία της πολιτικής συνοχή ω έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύη και ως βασικής επενδυτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ξεκάθαρη εδαφική διάσταση και πολύ βασική παράμετρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η πολιτική συνοχή φαίνεται στα αστικά κέντρα να επιτρέπει την ε, ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό μετά από μια δεκαετία εμπειρίας. Είναι πολλές οι χώρες που θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη στρατηγική προσοχή σε όλη την εφαρμογή της πολιτικής με συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις μεταρρύθμισης. Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ασχολείται με ζητήματα της κοινωνίας όπως η επασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η μετανάστευση, η παροχή ενέργειας, η βιωσιμότητα, η ανανέωση, αλλά δεν θα πρέπει να υπερφορτώσουμε και τη χάραξη πολιτικής ε, και να ε, είμαστε και έτοιμοι κάποιες φορές να ανταποκρινόμαστε και σε ανάγκες που προκύπτουν κατεπηγόντως. Θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι στις τρέχουσες πολιτικές συζητήσεις, αλλά να δούμε ξανά την διαχείριση και τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής. Η αρχή του management, της διαχείρισης, ε, πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους, γιατί ε, για την ώρα, εάν δεν την μελετήσουμε, θα συνεχίσει από κάποιους να θεωρείται προβολικά αυστηρή. Επίση, ο όγκο της νομοθεσίας ε, που σχετίζεται με την πολιτική συνοχή έχει γίνει αντικείμενο επικρίσεων. Χρειάζονται απλούστεροι και πιο ξεκάθαροι κανόνες, όπως ένας ενιαίο κανονισμό. Άμεση σχέση με όλα αυτά έχει και η, έχει και η ανάγκη για περισσότερη ευελιξία, εμέσω και αμέσω. Οι περισσότεροι από του εμπλεκόμενου σε αυτό το τομέα ζητούν μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορεί κανεί να δει πιο εύκολα τι ε, επερχόμενε εξελίξει και να ετοιμαστεί για να αντιδράσει γι' αυτό, όπω το απόθεμα για την ευελιξία, το περιθώριο για την ευελιξία. Επίση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικέ καταστάσει που επικρατούν σε διαφορετικέ χώρε. Ω προ του θεματικού στόχου, αυτό έχει να κάνει και με την ευελιξία, αλλά και με ένα άλλο θεμελιώδε ερώτημα. Δηλαδή, ποιοι είναι οι τομεί στου οποίου θα πρέπει να επικεντρώνεται η πολιτική συνοχή και πώ θα πρέπει οι θεματικέ ενότητε αυτέ να ε, γίνουν κατανοητέ στην πράξη. Εδώ είναι διαφορετικές οι θέσεις και η κατάσταση των διαφορετικών χωρών. Κάποιοι θέλουν την επικέντρωση της πολιτικής συνοχής σε κάποιους βασικούς στόχους με περισσότερη θεματική συγκέντρωση και περισσότερη ελαστικότητα. Χρειάζονται πραγματικές σχέσεις συνεργασίας και πραγματική συμπληρωματικότητα μεταξύ αυτών των κονδυλίων της συνοχής και άλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περισσότερο συνεκτικούς κανόνες λόγου χάρη. Όταν δει κανεί ένα κλασικό παράδειγμα από τις κλασικές παραμέτρους της αστικής διάσταση, αυτό ήταν ένα καυτό θέμα της επικαιρότητα και στις συζητήσει για το τελευταίο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τη χάραξη πολιτικής συνοχή. Αυτό θα συνεχιστεί και τώρα. Όπως το δίκτυο Γερμανίας-Αυστρίας αστικών κέντρων έχει δείξει, Το πού θα αποδοθούν τα κονδύλια ε, εξαρτάται από τις διάφορες προκλήσεις που προκύπτουν. Την ενεργειακή απόδοση, τις κλιματικές αλλαγές, την ε, ε, μετανάστευση, την ανανέωση και ανάπλαση που πολλές φορές χρειάζεται. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και οι νομικές βάσεις λίγο πιο ευέλικτε στη χρήση του. Η θεματική στόχη λόγου χάρη στην ε, θεματική ανάπτυξη στόχων είναι μια τέτοια, ένα τέτοιο παράδειγμα. Δεν χρειάζεται να είναι αυστηρέ οι διατάξει για να μπορούμε να προσαρμόσουμε του στόχου μα. Επίση, συχνά ε, συζητούμε και εδώ ε, και αλλού τι διασυνδέσει των αστικών κέντρων με την Ήπεθρο. Χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση των διασυνδέσεων αυτών. Καινοτόμε περιφερειακές πολιτικές μπορούν να σχεδιαστούν με θέματα όπως η κινητικότητα, η ενέργεια, ε, η παροχή, ο τουρισμός και η πρόληψη πλημμυρών. Εδώ η ευελιξία είναι ακρογωνιαίος λήθος του πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την αστική διάσταση. Λιγότερο διοικητικό άρθρος, λιγότερος φόρτος γραφειοκρατικός. Ως προς τη διαχείριση, η πλήρης εφαρμογή των αρχών εταιρικών σχέσεων είναι κάτι το σημαντικό. Είναι πολλοί εταίροι και ενδιαφερόμενοι που προτείνουν να εφαρμοστούν οι δεσμευτικέ διατάξει των εταιρικών σχέσεων βάσει του κανονισμού και όχι ο σημερινό κώδικα συμπεριφορά, λόγω χάρη. Επιτρέψτε μου να περάσω σε κάποιες από τις προκλήσεις, που, από τις συστάσεις μάλλον που τώρα έχουν εκφραστεί στο πρώτο πρόγραμμα δράσης των εταιρικών σχέσεων όσων εργάζονται υπό την αιγίδα αυτού του δικτύου αστικών κέντρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εταιρικέ σχέσει, ασχολούνται με τη διατύπωση συγκεκριμένων αξιολογήσεων και δράσεων για ζητήματα, τα οποία έχουν μια μεγάλη αστική διάσταση. Τέτοια ζητήματα Απλώς είναι προέκταση παλιότερων εταιρικών σχέσεων που ήδη έχουν εφαρμόσει το πρώτο πρόγραμμα δράσης τους. Κάποια άλλα αστικά κέντρα θα υποβάλουν το πρόγραμμα δράση του ε, στο εγγύ μέλλον δεύτερη και τρίτη γενιά και θα τα υποβάλουν και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο εντό του 2018 και 2019 Αυτά τα προγράμματα πρόκειται να ε, υποβληθούν. Η καταπολέμηση τη φτώχεια, το πρώτο πρόγραμμα δράση, η πρώτη εταιρική σχέση που ξεκίνησε το 2016 βάσει του Συμφώνου του Άμστερνταμ, αναφέρονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με, τις, ε, με τη διαρθρωτική αντιμετώπιση τη ε, φτώχεια μέσω τη πολιτική γειτονία και λύσει που πρέπει να προταθούν βάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Υπό αυτή την έννοια, η εταιρική αυτή σχέση καταπολέμηση τη φτώχεια επικεντρώνεται και σε σε ε, αντιμετώπιση του θέματος επίπεδο πολιτών αλλά και των αστικών κέντρων, ε, αναβάθμιση συγκεκριμένων γειτονιών λόγω χάρη αλλά και ένταξη των ανθρώπων ε, ανάλογα με την κατοικία τους στην πολιτική αυτή. Η χωρική συγκέντρωση, η εδαφική συγκέντρωση και εντοπισμός της φτώχειας σε συγκεκριμένες υποβαθμισμένες γειτονιές είναι ας πούμε ένα μέρος τη εταιρική σχέση που προτάθηκε με ανάπλαση κάποιων περιοχών σε αστικά κέντρα και ένταξη στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού τη συνοχής έχουν Έχει να κάνει με ανεργία, με ε, ανθρώπους που δεν έχουν τα διάφορα εκπαιδευτικά προσόντα, με ε, χαμηλά, χαμηλές ε, βιωτικές συνθήκες και το υποβαθμισμένο κοινωνικό ιστορικό. Εμπλέκονται διάφοροι εταίροι από διαφορετικά επίπεδα αλλά και ε, κάτοικοι από τις συγκεκριμένε περιοχές όπως προτείνει η εταιρική σχέση. Έτσι, η αστική ε, εδαφική στόχη είναι κάτι από αυτά που προτείνει η εταιρική σχέση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των υποβαθμισμένων περιοχών. Χρειάζονται ολοκληρωμένες στρατηγικές για να μην υπάρξει κατακαιρματισμός των κονδυλίων όπως αποδίδονται και να αξιοποιηθούν όλα αυτά τα χρήματα για την ανάπλαση αυτών των αστικών περιοχών προς όφελος και των συγκεκριμένων κατοίκων τους και άλλων πολιτών. Επίση, θα πρέπει τα κατημέλη στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση να συνσχεδιάσουν την καταπολέμηση τη φτώχεια και τη σχετική εταιρική σχέση με άλλου ε, κρατικού φορεί, με συνεργασία των κατοίκων και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Τώρα, η ένταξη των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία, άλλη εταιρική σχέση. Η εταιρική αυτή σχέση πρότεινε δύο συγκεκριμένε δράσει. Πρώτα απ' όλα, να δώσει τη δυνατότητα ανάμειξη ε, κάποιων στρατηγικών στα αστικά κέντρα μέσω ε, δανείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη των μεταναστών μπορούν να συνδυαστούν καλύτερα με τα κονδύλια από τα διευθυντικά, από τα ε, ταμεία συνοχής και από την ΕΤΕ. Προβλέπεται καλύτερη και αμεσότερη πρόσβαση στα, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ένταξης και στις πόλεις πλέον οι δημοσιονομικές γραμμές για την ένταξη μέσω των Ταμείων Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Ταμείων Συνοχής, των Διευθυντικών Ταμείων μπορούν να ε, συνδυαστούν αρκεί να υπάρξει αρκετό συντονισμό σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των διαφορών υπουργείων, πράγμα που τώρα δεν υπάρχει. Ε, τα χρονικά περιθώρια ε, με τον καθορισμό προτεραιοτήτων, αιρεσιμότητα ε, κανόνων για την υποβολή εκθέσεων είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ του προ στιγμή. Παρόλο που ο στόχο είναι χονδρικά κοινό, η ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην κοινωνία. Χρειάζεται λοιπόν μια ομαλή ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στον κοινωνικό μας ιστό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια για την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση Ένταξης εντός και σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Τρίτη εταιρική σχέση. Αυτή που έχει να κάνει με την αστική κινητικότητα. Η εταιρική αυτή σχέση δείχνει την ανάγκη να υπάρχουν βιώσιμα προγράμματα για την αστική κινητικότητα με τα κατάλληλα ποσά για να υποστηρίξουμε τη διάσταση αυτή και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Η εταιρική αυτή σχέση προτείνει τα, ε, οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκησης, πόλει και περιφέρειες να εμπλέκονται περισσότερο στον ε, πολιετή δημοσιονομικό προγραμματισμό. Η αστική κινητικότητα καλεί τι αστικέ και δημοτικέ αρχέ να, να συμμετέχουν άμεσα στον καθορισμό θεματικών προτεραιοτήτων και εργαλείων για την υποστήριξη των σχετικών εξελίξεων. Ο κώδικα συμπεριφορά τη εταιρική σχέση και αυτή η αρχή πρέπει να ενταχθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής με μια εξάντερη για την πλήρη εκδίπλωση των δυνατοτήτων της εταιρικής αυτής σχέσης. Να πάω τώρα στην τελευταία από τις τέσσερις εταιρικέ σχέσεις, ε, την ε, κυκλική οικονομία και τη σχετική εταιρική σχέση που αναφερθήκε προηγουμένως σήμερα το πρωί. Για τη διαχείριση αυτής της εταιρική σχέσης χρειάζεται συμμετοχή ε, περιφερειών, αστικών κέντρων και υπαίθρου και η συμμετοχή των φορέων. Η εταιρική αυτή σχέση είναι, είναι σημαντική για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα αστικά κέντρα. Και μετά το 2020 χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. επίκεντρο της εταιρικής αυτής σχέσης είναι ότι η πολιτική συνοχή πρέπει να επιτρέπει την ε, ε, ανανέωση και την ε, ανάπτυξη σε επίπεδο υπαίθρου και αστικών κέντρων με σχέσεις συνεργασίας, με την κατάλληλη ατζέντα, με εταιρικέ σχέσεις και κοινοτόμες δράσεις σε αστικά κέντρα και υπαίθρου. Η αστική ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα συνεργαστικό πείραμα που ξεκίνησε το 2016 και κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί και μετά το 2020. Είναι σημαντικό για την περαιτέρω εξέλιξη και ε, υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης αυτών των εταιρικών σχέσεων να υπάρχει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και με το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, η φάση απαντήσεων και αντιδράσεων στην μέχρι τώρα εφαρμογή των προγραμμάτων δράση θα αρχίσει σύντομα με τη συμμετοχή των πολιτικών θυνόντων, των ενδιαφερομένων που ελπίζουμε να συνεισφέρουν για να επηρεάσουν την σύνταξη συστάσεων για το δεύτερο μέρος της χρονιάς φέτος με τη δεύτερη και τρίτη γενιά των εταιρικών σχέσεων που έρχονται. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν και μέσω ενός ιστοτόπου που υπάρχει η διεύθυνσή του στις διαφάνειες και με φυλάδια. Η πρόθεση της αστικής ατζέντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να ε, εφαρμόσουμε τις αρχές της καλύτερης νομοθεσίας, καλύτερης ρύθμισης και καλύτερης γνώσης και να τα εντάξουμε στις εταιρικές μας σχέσεις. Ελπίζουμε και στην επόμενη γενιά να είμαστε εδώ για να σα παρουσιάσουμε τα πορίσματα αυτών των περιοδικών σχέσεων και μην διστάσετε για τι ερωτήσει. Γενικό Σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομική Ανάπτυξη τη Πολωνία. Το θέμα είναι ή σε διδάγματα που αντιλήθηκαν στην Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είναι κάπως πολύπλοκος ο τίτλος, αλλά θα προσπαθήσω ουσιαστικά να συμπληρώσω τα όσα Συμφωνώ σε πολλά όπως είπαν οι συνάδελφοί μου, αλλά θα ήθελα να προσθέσω στις απόψεις τους κάποιες ε, ε, ακόμη σκέψεις μου. Ποιο είναι στην αστική, στις περιοχές, στην Ήπεθρο, στις τα κτλ. Πρέπει να βρούμε μια κοινή προσέγγιση για όλες αυτές τις περιοχές. Εγώ λοιπόν μιλώ κυρίως για εδαφικές πολιτικές και όχι για αστικές, αγροτικές ε, ή περιφερειακές. ο καθηγητής επηρεάζουν επικοινωτρόπως ε, και σημαντικά τις προοπτικές και την ποιότητα ζωής των πολιτών ανάλογα με το που ζουν. Επίσης, επηρεάζουν επικοινωτρόπως ε, και σημαντικά τις προοπτικές και την ποιότητα ζωής των πολιτών ανάλογα με το που ζουν. Επίσης, είναι προφανές και το βλέπετε και στα έγγραφα της Κομισιόν, παραδείγματος χάρη από το 2017, σε σχέση μόνο με την πολιτική συνοχή αλλά και με την παγκοσμιοποίηση, τα κοινωνικά θέματα, το μελλοντικό προϋπολογισμό. Όλα αυτά τα έγγραφα υπογραμμίζουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη και πεδίο για εδαφική πολιτική σε ευρωπαϊκό, εθνικό πιο αποτελεσματικές θα είναι οι δημοσίε πολιτικέ σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο αν λάβουν υπόψη τα θετικά στοιχεία και όχι μόνο τα αρνητικά να τα βλέπουν συνολικότερα από την αδαφική τους σκοπιά και όχι την τοπική. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα Τις πανέρθα εδώ για να πω ότι σήμερα η πολιτική συνοχής δεν έχει, ο έδαφος επηρεάζεται και διαφορετικά η κατάσταση στη περιφέρεια. Αλλά τι μπορεί να κάνει η πολιτική συνοχή. Δεν έχει ξοποιήσει το πλήρες δυναμικό ώστε να βοηθήσει όλα τα είδη δαφών. Η υποβάθμιση του ρόλου της ε, πολιτικής συνοχής, έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνονται ορισμένοι και αυτό το βλέπουν. Επίσης έχουμε το προσανατολισμένη εφαρμογή συντονισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που λείπει. Τώρα όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από την πολωνική συντονισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που λείπει. Τώρα όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι από την πολωνική οπτική γωνία η πολιτική συνοχή ε, τα καταφέρνει παρόλα αυτά ολοκληρώσαμε την ε, επιβεβαιώνει ότι πολιτική συνοχής έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να πετύχει σύγκληση στις χώρες και στις περιφέρειές τους. Αυξάνει επίσης την ανταγωνιστικό αύξηση κεφαλαίου, μείωση φτώχειας, οικονομική άνθηση των μεγάλων ιδιοσπόλεων, οικοδόμηση δικτύων, συνδεδεμένων δικτύων μεταφορών κτλ. Αν δείτε πιο κοντά και το σύστημα του earmarking, μας βοηθάει να βάλουμε προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την παροχή υποστήριξη σε project και περιοχέ ε, Ευρωπαϊκή Προστέμενη αξίας, σε ό,τι αφορά το σύστημα τη αρισιμότητα ε, μεταξύ των διαφόρων τμήματων τη διακυβέρνηση. Υπάρχουν εδαφικά εργαλεία που έχουν πολύ καλή επίδοση στις διάφορες ε, πτυχές της συνεργασίας και του συντονισμού. Δεν μπορούν όμως όλα να προκαλέσουν τις απαιτούμενες αλλαγές και να βοηθήσουν όλα τα εδάφη και όλες τις περιφέρειες να ξεδιπλώσουν το όμως δεν μπορούν όλα αυτά μαζί να περκεράσουν ε, τις επίμονες αυτές διαφορές και προβλήματα. Για παράδειγμα τους χάρη, λόγω της βοήθειας αυτής, βελτίωση της προσβασιμότητας, αύξηση των περιφερειών, αλλά ταυτόχρονα επιμένουν οι ανισότητες αύξηση των ε, περιφερειακών ή υποπεριφερειακών ανισοτήτων ε, συγγνώμη για το χάρτη που δεν τον βλέπετε καλά, αλλά στο υποπεριφερειακό επίπεδο βλέπουμε να εμένουν κάποια προβλήματα ή μάλιστα ακόμη να μεγεθύνονται σε κάποιες περιπτώσεις. Και δύο είναι αυτοί που χάνουν περισσότερο, αν μπορώ να το πω έτσι. Η μεσαίο μεγέθους πόλης και η ύπεθρος, οι αγροτικές περιοχές που απειλούνται από μόνιμη περιθωριοποίηση. Αυτή η εικόνα όμως δεν σχετίζεται με την ιστορία, τουλάχιστον όχι όσο στενά θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, ε, οι δύο πόλοι Δύση Ανατολή, όχι, είναι πολύπλοκα τα πράγματα σήμερα και έχουν να κάνουν ε, με τις περιφέρειες. Σε το και εγκομιάζουμε την ε, πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε προβλήματα, έχουμε μεγάλες ανισότητες, συγκέντρωση των ευκαιριών σε περιορισμένε περιοχέ. Και αυτές οι περιοχές μειώνονται ακόμη περισσότερο. Άρα, κοινή αγορά, ε, παγκοσμιοποίηση ε, είναι ισχυρές, επηρεάζουν και δεν μπορεί η πολιτική συνεχίσει να αναστρέψει την κατάσταση εντελώς. Ταυτόχρονα σε περιοχών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αυτό θα μπορούσε να μα κάνει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά, όχι μόνο τα χρήματα, οι πολιτικέ συνοχίζεται κατάλληλα με εθνικέ, περιφερειακέ και τοπικέ πολιτικέ. Ωραία το λέει κανεί, αλλά τι εκτόμιο κατάλογο με αυτόν που παρουσίασε ο Ανδρέα Πόσε. Αλλά από την πολιτική πολωνική σκοπιά ποιοι είναι οι παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν. ένα μηχανισμό συντονισμού μεταξύ των διαφόρων τομεακών μέσων που θα λαμβάνει υπόψη την εδαφική διάσταση. Εστίαση ε, στην επίτευξη μεταξύ των προγραμματών που χρηματοδοτούνται από την πολιτική και τα οποία εφαρμόζουμε. Και αυτά τα προγράμματα εν μέρη μόνο έχουν εκπληρώσει ε, τα, τους στόχους. Επίσης, πρέπει να δώσουμε κίνητρα και στους κοινωνικούς εταίρους με εστίαση στους εταίρους και στη συγκεκριμένη περιοχή. Επίσης θα πρέπει να υλοποιήσουμε με αποτελεσματική πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και ένα περιβάλλον πειραματισμού. Γιατί η αποκέντρωση έφερε πραγματικά μεγάλη εφευρετικότητα. Οι πολιτικέ περιφέρειες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με πολλά ακόμα το θέμα αυτό που δεν μπορώ να σας παρουσιάσω ε, συγκεκριμένα τα πορίσματα, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα έγγραφο στη σύνταξη του οποίου με τον Τζον Μπάτλερ, τον Γιακίμ Ολιβέηρα Μάρτιν και τον Πίτερ Βόσνερ ε, συνέταξε το 2017 το Πασίσμα για το τι πρέπει να αλλάξει. Αρχής γενομένης από τη στρατηγική προσέγγιση. Θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική εάν είναι στο κέντρο των στόχων ε, των στρατηγικών για την Ένωση μετά το 2020. Είναι αυτή η στρατηγική πολύ τους αναγκαία. Χωρίς την πολιτική συνοχή θα είναι μία απλά στρατηγική σαν όλες τις άλλες και δεν θα είναι μια στρατηγική που θα καταστήσει σημαντική την ε, εδαφική διάσταση και την πολιτική συνοχή. Εν συντομία κάποια άλλα, φυσικά αυτό πρέπει να χώρα. Ποιος είναι ο τους. Και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις διάφορες πολιτικές κτλ. κτλ. Όμως θα πρέπει στα σαν να ε, εστιάζουν στις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις για είναι λογικό. Και άλλες πολλές είναι οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει που τις βλέπετε συνοπτικά σε αυτή τη διαφάνεια. Και είναι και κατά πολύ παρόμοιες με αυτές που ανέφερε ο Αντρέας και δεν θέλω να τις ε, απαριθμίσω εφόσον τελειώνει ο χρόνος μου και δεν θέλω. Έχει τον τίτλο 7η έκθεση συνοχής. Πρέπει να σας πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένος. Γιατί οι προτάσεις ε, αυτής της έκθεσης εστιάζουν κυρίως στην εκτέλεση για να το θέσω έτσι. Στην έκθεση συνοχής ε, υπάρχει γιατί τελικά φέρνει δυσκολίες. Μόνο αν έχουμε μια νέα πλατφόρμα προγραμματισμού ε, και δέσμη μέτρων. Επίσης θα πρέπει η ανάλογα με τις εδαφικές ανάγκες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ναι, να διατηρήσουμε δηλαδή την ευρωπαϊκή αξία, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αυτό το συνδυασμό των διαφόρων μέτρων για να είναι προσαρμοσμένα στο τοπικό επίπεδο και τέλος η χρήση των αποθέσεων. Είχαμε εδώ μια εθνική προσέγγιση ε, την άποψη του μεγαλύτερου δικαιούχου από το Ταμείο Πολιτικής Συνοχής σε ζητήματα ευρωπαϊκών υποθέσεων της ε, ε περιφέρειας της Ile de France στη Γαλλία θα μας κάνει μια παρουσίαση θα μας πει λοιπόν να μας δώσει στοιχεία από το τι γίνεται επί τόπου feedback from the ground για μια πιο απλή και αποτελεσματική ευχαριστώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για την ε, υποδοχή σας αλλά να ευχαριστώ και τον Μάρκ Ζουλό τον ε, εισηγητή της έκθεσης για την πρόσκλησή του καλωσορίζω, μάλλον χαιρετίζω και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως τους Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα να κάνω πρώτα μια διαπίστωση. Η περιοχή Ile de France είναι η πρώτη περιφέρεια της Γαλλίας 30% του ΑΕΠ, 20% του πληθυσμού, ο μεγαλύτερος πόλος οικονομικής ανάπτυξης και ο πρώτος ακαδημαϊκός πόλος. Είναι και από τις πιο πλούσιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, παρά αυτά τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, στη Γαλλία, στην Ile de France, υπάρχουν πολύ μεγάλες εδαφικές αποκλίσεις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές, ε, υποπεριφερειακές λοιπόν αποκλίσεις. Υπάρχουν μάλιστα πραγματικοί θύλακες φτώχειας. Ε, η περιοχή, το διαμέρισμα του Σεν Σαντονί ε, είναι από τις πιο φτωχές ε, τα πιο, πιο φτωχά διαμέρισματα της Γαλλίας. Το 70% του εδάφους της περιφέρειας αυτής είναι γεωργικό και χρειάζεται συγκεκριμένη ε, έχει συγκεκριμένε ανάγκε για να μπορέσει να εξασφαλίσει βιώσιμη γεωργία. Επίση, η περιοχή τη Ile de France δεσμεύεται έτσι ώστε το αστικό σκέλος ε, του εδάφου να παραμείνει ελκυστικό. Και γι' αυτό βεβαίω έχουμε πραγματογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τον ε, αστικό άξονα, μια και ο αστικό άξονα τη περιφερειακή πολιτική αποτελεί περίπου 20% του επιχειρησιακού περιφερειακού μας προγράμματος. 112,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία κατανέμονται ε, σε 15 ε, προγράμματα ε, ET συγκεκριμένοι φάκελοι λοιπόν συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που αφορούν αυτά τα αστικά εδάφη τις αστικές περιοχές έχουμε λοιπόν πολλαπλά ταμεία τα οποία υποστηρίζουν αυτά τα project υπάρχει μεγάλη, μεγάλη υποστήριξη στα προγράμματα αυτά ε, από το Κοινωνικό Ταμείο, από το ΦΕΝΤΕΡ. Ε, θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε μια σειρά από για την περίοδο 2014-2020. Για πρώτη φορά η περιοχή της Ile de France, όπως όλες οι περιφέρειες, είναι πλέον η αρχή διαχείρισης των ε, χρημάτων αυτών. 540 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΕΝΤΕΡ, το ΦΕΑΝΤΕΡ, το Κοινωνικό Ταμείο 185,4 εκατομμύρια ευρώ από το ΦΕΝΤΕΡ, 672 εκατομμύρια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, μεταξύ του κράτους και της περιφέρειας, εκεί υπάρχει κατανέμιση και και 375 εκατομμύρια σε ό,τι αφορά το σκέλος απασχόλησης και ένταξης. Και υπάρχει και ένα άλλο κονδύλιο, λίγο λιγότερο από 60 εκατομμύρια ευρώ, από το ΦΕΑΝΤΕΡ. Από το 2016 μετά την αλλαγή ε, της ε, διακυβέρνησης της περιφέρειας υπάρχει μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ε, που θέλουμε να είναι φιλόδοξη και η οποία αποτελείται από τέσσερις άξονες. Θα αναφερθώ λίγο σχετικά διότι η πολιτική συνοχή ε, είναι κεντρική σε αυτό το εγχείρημα. Ο πρώτος άξονας είναι να είμαστε παραδειγματικοί ε, στην χρήση και την κατανάλωση των ευρωπαϊκών ταμείων. Θα μου πείτε εννοείται. Εννοείται αλλά καλό είναι να το λέμε κιόλας ε, διότι δεν ήταν πάντα έτσι στο παρελθόν. Δεύτερος άξονας, να συνοδεύσουμε καλύτερα τους ε, εμπνευστές των project. Τρίτος άξονας, να υπάρχει μια στρατηγική αποκεντρωμένη συνεργασίας και τέταρτο άξονα ε, να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό που να επιτρέπει να ενημερώνεται το ευρύ κοινό για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ για να ε, μπορέσει η δράση αυτή να είναι εκτιμητέα. Θα πρέπει επίση να γίνουν μελέτε ε, που θα φωτίζουν στοιχεία γύρω από τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ στο έδαφο τη Ile de France για να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε την συνεισφορά την ευρωπαϊκή στις δραστηριότητε τοπικές και αυτή είναι η καρδιά της παρέμβασής μου σήμερα ε, για να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε τη χρήση αυτών των ταμείων για πρώτη φορά η περιφέρεια το Μάιο και Ιούνιο του 2017 ε, οργάνωσε μια διαβούλευση διαβούλευση με 70 ε, χρήστες project, 100 ε, άτομα περίπου συνολικά εμπλεκόμενων φορέων, ε, δικαιούχων ε, των project αυτών, ε, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από άτομα που έχουν διαφορετικό νομικό καθεστώς, δηλαδή μιλήσαμε και με ενώσεις και με τοπικές αρχές και με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με πόλεις ανταγωνιστικότητας και με κοινωνικούς φορείς. Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν διαφορετικά ταμεία, όλοι αυτοί έχουν διαφορετικές θεματικές, διαφορετικά προβλήματα και όλοι έχουν εμπειρία πολύτιμη για την αρχή διαχείρισης αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος ήταν ε, βέβαια να μπορέσουμε να συλλέξουμε τις ε, εμπειρίες τους αλλά και το τι είχαν να μας πούν για τη χρησιμοποίηση αυτών των ταμείων και να τους δώσουμε βέβαια τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις όταν ξεκινεί, ξεκινάει πλέον η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής έτσι ώστε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα αυτής της πολιτικής και την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τους δημόσιους λειτουργούς, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε ε, τη φωνή των βασικών δικαιούχων ε, τους ανθρώπους αυτούς για τους οποίους ε, λαμβάνουν χώρα αυτές τις πολιτικές. Να δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία. Βεβαίως έχουμε στη διάθεσή σας ε, ε, εδώ σε εσά τους ευρωβουλευτές και για όποιον άλλο να ενδιαφέρεται έχουμε τα πλήρη στοιχεία και τις εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει έχουμε περίπου 100 φάκελους στη διάθεσή σας σήμερα μπορείτε να τα παραλάβετε κάποια στοιχεία θα σας δώσω λοιπόν τα οποία είναι αρκετά αποκαλυπτικά σε ό,τι αφορά τη σημασία των διαθροτικών ταμείων ε, για αυτά τα project τα οποία ε, είναι προς όφελος ε, των κατοίκων της περιοχής. Καταρχήν 8 στους 10 συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι από την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά αυτά κονδύλια. 64% εξ αυτών μας είπαν ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία συμμετέχουν σε μία δημιουργία ε, ενός ε, συναισθήματος ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Πολύ καλό αποτέλεσμα αυτό. Δείχνει λοιπόν ότι αυτό το, αυτό το αίσθημα του ανήκειν ε, στο ευρωπαϊκό σχέδιο συνδέεται με τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά ταμεία. Από την άλλη βέβαια, όπως συχνά έχουμε ακούσει και ελέγχθηκε εδώ, οι συμμετέχοντες στα project έχουν εντοπίσει μια σειρά από εμπόδια που ορισμένες φορές ε, πραγματικά ε, μπλοκάρουν την ολοκλήρωση των project ε, και τελικά καταλήγουν να είναι αντιπαραγωγικά. Ένα στου δέκα μας λέει ότι 30% του χρόνου του τον σπαταλά για τι δύο του υποχρεώσεις αντί να ασχολείται με το project του. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται οπωσδήποτε απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών ένα άλλο διοικητικό εμπόδιο. Μόλις 13% των απάντησαν θεωρούν ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία ε, οδηγούν στο να επιτευχθεί ο στόχος τους πιο γρήγορα. Γι' αυτό λοιπόν έχει δημιουργηθεί μια ομάδα ατόμων υποστήριξης που να βοηθούν στην ανάπτυξη του project. Δεν θέλουμε απλώς εμείς να κατηγορήσουμε το πώς έχει δομηθεί αυτή η πολιτική συνοχή. Ε, θέλουμε κατά την εφαρμογή να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα, διότι έχουμε και εμεί ευθύνη. Αναλαμβάνουμε λοιπόν ευθύνη, την ευθύνη αυτή, προσπαθούμε ε, να οδηγήσουμε σε μια πιο ε, εύρυθμη ροή τη εφαρμογή. Έχουμε λοιπόν μια ομάδα ατόμων που διευκολύνουν, που βοηθούν του ε, συμμετέχοντες στα project να επιταχυνθούν, επιταχυνθεί η διαχείριση διαφόρων project, ο καθένα να έχει ένα συνομιλητή που να τον βοηθάει από την αρχή μέχρι το τέλο αυτή η διαδικασία ε, κατέστη εφικτή διότι πέρασαμε από 21 υπαλλήλους στους 54 σε αυτή την ομάδα που βοηθούν λοιπόν ε, όσους προωθούν τα project. Θέλουμε έτσι να μπορέσουμε να διαφημίσουμε ε, τα ευρωπαϊκά κοινωνικά ταμεία, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτές οι δυσκολίες θεωρούνται, ε, θεωρείται ότι μπορούν να ξεπεραστούν. Αυτό λέει το 70% από κόστος. Ε, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τάση. Δεύτερο, να μειώσουμε τον αριθμό των δικτών και να, τις προσ, να προσαρμόσουμε στις τοπικόστος. Ε, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η τάση. Δεύτερον, να μειώσουμε τον αριθμό των δικτών και να τις να τους προσαρμόσουμε στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Και αυτό ελέγχθη πολλάκι σήμερα το πρωί. Τρίτον, τα επιχειρησιακά προγράμματα να είναι πιο ευέλικτα, να μπορούν να προσαρμόζονται στο χρόνο και στις εξελίξεις, σε τοπικό επίπεδο. Ζούμε σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει μια επιτάχυνση. Κάτι δηλαδή που ίσχυε το 2014 μπορεί να μείνει και στις εξελίξεις, σε τοπικό επίπεδο. Ζούμε σε ένα πλαίσιο όπου υπάρχει μια επιτάχυνση. Κάτι δηλαδή που ίσχυε το 2014 μπορεί να μην ισχύει σήμερα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη πέρα από τις πολιτικές διακυμάνσεις, τις πολιτικές εξελίξεις, αυτές, ε, αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να καταστούν πιο ευέλικτα. Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε σε κάποιες θεματικές, ε, σε ε, συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία θα είναι πιο ορατά ε, θα, μια, θα υπάρχει μια μαζική ε, έκθεση σε αυτά τα προγράμματα, ε, μειωθούν οι έλεγχοι. Είναι απαραίτητη η έλεγχη βέβαια, αλλά θέλουμε να, έχουμε, να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνη μεταξύ όσων τρέχουν τα project, των τοπικών αρχών και των ευρωπαϊκών αρχών για να μειωθεί έτσι και ο αριθμός των ελέγχων. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 και 6 ελέγχους ορισμένες φορές για ένα και μόνο project. Και βέβαια είναι και επιζήμιο στην σχέση που θέλουμε να έχουμε και να δημιουργήσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε λοιπόν ένα συγκεκριμένο μέτρο για να υπάρξει απλοποίηση. Τη θέσπιση μιας αρχής ε, label, περίοδο, πραγματική περίοδο, ε, να έχουν αυτό το σήμα της αξιοπιστίας και να ελέγχονται λιγότερο. Βεβαίω οι έλεγχοι χρειάζονται. Μιλάμε για δημόσια κονδύλια, δημόσια χρήματα. Αλλά μπορούμε να καταστήσουμε αυτούς τους ελέγχους ε, ε, λιγότερο ε, προτείνουμε αυτό το μέτρο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, αυτά τα εμπόδια στα οποία αναφέρθηκαν όσοι συμμετέχουν στα project. Έχουμε και μια σειρά από παραδείγματα τα οποία θα βρείτε στις εκθέσεις μας. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία ζητούνται από τους συμμετέχοντες. Αυτό το λένε πολλοί στη διαβούλευση. Και αυτά τα δεδομένα, εφόσον δεν είναι ενημερωμένα, ε, μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν θα χρηματοδοτηθεί το project. Ε, και αυτό τελικά είναι εντελώ παραγωγικό και για την αρχή διαχείρισης, αλλά και 12 ακόμα δείκτες ε, για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Σε ό,τι αφορά, όχι μόνο λοιπόν αυτοί οι δείκτες είναι πολλοί, αλλά αυτή καθ' αυτοί ορισμένες φορέ, διότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι εγκαταλείπουν ε, την, το πρόβλημα ε, στόχο να βοηθήσουμε τους άστεγους. Ε, αλλά για να συμπληρωθεί ο φάκελος ζητούμε τη διεύθυνση των ανθρώπων αυτών που είναι άστεγοι. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ μιλάμε για θέατρο του παραλόγου. υπάρχουν τα κριτήρια τα οποία δεν είναι έτσι και τόσο ευχάριστα project, ε, έτοιμα μάλλον για project ε, ε, να βοηθούν γυναίκες που έχουν υποστεί ενδοχογενειακή βία. Ε, θέλουμε να απομακρύνουμε αυτές τις γυναίκες από τον, την πηγή κινδύνου, να μην είναι γνωστή η διεύθυνση, αλλά παρόλα αυτά ζει κατάρτιση ανθρώπων που έχουν προβλήματα με τη δικαιοσύνη και εκεί υπάρχουν παρεμφερεί ζητήματα. Τελειώνοντας, ε, να υπογραμμίσω τις τρεις βασικές δεσμεύσεις της περιφέρειας Ile de France ε, στα πλαίσια αυτής της συζήτησης που γίνεται για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Πρώτον, ΔΕΡ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης πρέπει να ελαφρυνθούν, να μειωθούν οι έλεγχοι, να είναι πιο ευέλικτη η εφαρμογή και να, μια, να συγκεντρωθούμε θεματικά στις ε, προσδοκίες όσων υποβάλλουν τα project. Επίση πρέπει να υπάρχει αυτό το, αυτό το labeling, οι κυρίε βουλευτέ. Η πολιτική συνοχή είναι η ψυχή του ευρωπαϊκού σχεδίου και τη ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Κάθε μέρα αποδεικνύει στα εδάφη τη Ένωση ότι έρχεται να καλύψει σημαντικέ ανάγκε των εδαφών και των Ευρωπαίων πολιτών. Και το γεγονό ότι Υπάρχει βεβαίω πέρσι ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την ύπαρξη της πολιτικής αυτής. Ανταποκρίνεται σε ανάγκε μιας Ευρώπης που θέλουμε να οικοδομήσουμε, μια συγκεκριμένη Ευρώπη που να ενσαρκώνεται ε, στα εδάφια αυτή. Η, περιοχή Λιντεφρόντ όχι μόνο είναι έτοιμη, αλλά είναι και αποφασισμένη να σα συνοδεύσει, κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, στην προσπάθεια αυτή για να οικοδομήσουμε αυτή τη νέα Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστούμε για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ευχαριστούμε και για την ε, γραπτή δήλωση που λάβαμε από την περιοχή Φράνς για το μέλλον της ε, περιοχής και γενικώ της πολιτικής συνοχής. Σας ε, ευχαριστούμε, θα διαφωτίσει και τις σημερινές μας συζητήσεις. Ανοίγω λοιπόν τώρα το βήμα στους συναδέλφους της Επιτροπής Ρέμπη. Ποιος θα ξεκινήσει, δεν έχω ακόμη κατάλογο γορτών. Ο κύριος Φανίστελ Ρόι. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι κανείς σε πειρασμό να μπει σε λεπτομέρειες σε σχέση με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπατε ή να πάει απευθείας σε βιαστικά συμπεράσματα, διότι φέτος ήδη μας απασχολεί το τι θα γίνει με το μέλλον των δημοσιονομικών προοπτικών και το τι αποφάσεις πρέπει να λάβουμε. Έχω λοιπόν μια ερώτηση προς τον καθηγητή Ροντρίγκερ. στην κατηγοριοποίηση των ε, περιοχών ε, και περιφερειών της Ευρώπης ως τώρα έχουμε τις λιγότερο και περισσότερο αναπτυγμένες. Εσείς έχετε μια άλλη οπτική γωνία για να εξετάσετε το θέμα του εισοδήματος και είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβω εγώ, διότι είναι ένας εντελώς τρόπος προσέγγισης της όλης συζήτησης, όχι πια με το ΑΕΠ και με διαφορετικά κριτήρια κατηγοριοποίησης. Ξέρετε βάσει των δικών σας γνώσεων, πώς θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να έχουμε καλύτερη ταξινόμηση για το επόμενο διάστημα, την επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Το ερωτώ και προς τους υπολείπους προσκεκλημένους. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να βρούμε καλύτερα κριτήρια, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε επιχειρησιακό λειτουργικό επίπεδο βλέπουμε να υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές ε, ανισότητες εντός των διαφορών περιφερειών. Και η άλλη μου ε, ερώτηση έχει να κάνει με όσα μας είπε κυρία ε, και σε σχέση με τη δήλωση της περιοχής Ile ε, εάν δείτε τι λένε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λένε ότι δεν έφερε αποτέλεσμα το, ε, ούτε το Κοινωνικό Ταμείο ούτε το Ταμείο της Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κι όμως στην πράξη θέλουμε κάποια μορφή συνεργασίας ώστε να μπορέσουν οι πόλεις, οι κοινωνικοί εταίροι να ε, συνδυάσουν τα κονδύλια και τις επενδύσεις από αυτά τα ταμεία. Η δήλωσή σας πάρα πολύ μου άρεσε αλλά μπορείτε ίσως να μου πείτε περισσότερα για να ενισχύσουμε και τα επιχειρήματά μας για την πολιτική συζήτηση που θα έρθει τους επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε. Κύριε Ζουλό, θέλετε το λόγο τώρα ή θέλετε να κάνετε τη σύνοψη της όλης συζήτηση στο τέλος. Όχι μόνο κοιτάζει να μειώσει τις ανισότητες, πράγμα που είναι και πρωταρχικός της στόχος, αλλά τρόπον την καταλάβουμε αυτή την ενδεχόμενη εγκατάλειψη και αυτό που μας είπατε εσείς για το κοινωνικό ταμείο και τη σημασία του. Ήθελα να μου πείτε πώς το βλέπετε κι εσείς από την οπτική γωνία του, ε, ε, της Ile της περιοχής σας. Κυρία Μπρέσο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις παρουσιάσεις τους που ήταν άκρος ενδιαφέρουσες. Γενικώ φαίνεται με διαφορετικούς τρόπους πως η πολιτική συνοχής κατά πάσα πιθανότητα θα μπορούσε να ε, εξελιχθεί σε πολιτική συνεχής και ανάπτυξης. Χρησιμοποίησαμε τον όρο ανταγωνιστικότητα που είναι σωστός, όμω το ιδανικό θα ήταν ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Διότι υπάρχει πρόβλημα στην Ευρώπη με τις περιοχές που έχουν χαμηλότερη ανάπτυξη και έχει να κάνει με αναδυόμενες χώρες και οικονομίες όπου αυτή τη στιγμή γίνονται επενδύσεις για την αναπτυξή τους. Οπότε έχουν το πλεονέκτημα να έχουν επενδύσεις βάσει των νέων τους. Οπότε έχουν το πλεονέκτημα να έχουν επενδύσει βάσει των νέων τρόπου του παρελθόντο και πρέπει να ανανεωθεί πλήρω. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη σε σχέση με άλλε περιοχέ του κόσμου, ε, για να μην πω με όλο τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό δεν αφορά μόνο τι περιοχέ που είναι λιγότερο αναπτυγμένε, ούτε τι περιοχέ με μέσο εισόδημα. Αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Εάν δούμε την έκθεση περί συνοχής, ε, είναι κάτι που είναι προφανέστατο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Προφανές είναι και, είναι και τα εξή διότι να Θα πρέπει από κοινού να συνδυάσουμε την πολιτική συνοχή και το πρόγραμμα Juncker για να βελτιώσουμε τη συνολική μας επενδυτική ικανότητα. Δεν θα πρέπει να είναι μία η παρέμβασή μας, αλλά να συνδυαστεί με πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ήθελα να κάνω μια η παρεμβαση μας αλλα να συνδυαστει με πολλα χρηματοδοτικα εργαλεια θελω να κανω μια ερωτηση για τις περιοχές που βρίσκονται στην παγίδα του μέσου εισοδήματο. Κάτι που, όπως είπε και ο εισηγητής μας, ο κ. Ζουλό, ε, δείχνει ποια είναι η βασική πρόκληση για τη νέα περίοδο προγραμματισμού. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ο καθηγητής Ροντρίγκε μας έδωσε κάποιες πρώτες ενδείξεις, πολύ ενδιαφέρουσες, και ήθελα να κάνω την εξής ε, σκέψη, το εξής σχόλιο. Ίσως το συνολικό σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να κοιτάξουμε προσοχή πράγματα που συνέβησαν στο πρόσφατο θα έλεγα παρελθόν της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή την τάση πολλών περιοχών και περιφερειών με χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης αντί να προβλέπουν νέες παραγωγικές δυνατότητες να προσελκύουν χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια επιχειρήσεις και εταιρείε στην επικράτειά τους ε, ε, κλέβοντάς τις από άλλες περιοχές. Στην ουσία δεν υπάρχει κέρδος εδώ. Δηλαδή Εάν ε, η εταιρεία που θα κλείσει στη δική σου γειτονιά έρθει στη δική μου, τελικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ίδιο θα συμβεί. Αλλά επίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν μια φτωχότερη χώρα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πράγματα εκεί είναι φθηνότερα, ε, θα φύγει από μένα εταιρεία και θα έρθει σε σένα. Ε, σε κάποιον άλλο τέλο πάντων, και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάπω έτσι ναρκώνεται και η αγορά. Έχουν προκύψει πολλέ τέτοιε περιπτώσει, ε, τι γνωρίζουμε πιστεύω και είναι ένα από τα σημεία όπου για το μέλλον θα χρειαστεί κάτι να κάνουμε. Έχουμε επιλύσει κάποια προβλήματα, προσωρινά ίσως, σε κάποιες περιοχές, δημιουργώντας όμως προβλήματα σε άλλες αντιστοίχω περιοχές, μέσω ενός ανταγωνισμού που είναι και αθέμητος αθέμητος γιατί βασίζεται στο χαμηλότερο δυνατό κόστος παραγωγής και μάλιστα με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να γίνουν μετακινήσεις επιχειρήσεων. Δεν είναι και πολύ θεμητό αυτό, έτσι. Και πολλές επιχειρήσεις τις χάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φρονώ λοιπόν ότι το θέμα αυτό πρέπει να εξεταστεί και να δοθεί προσοχή Πολλές πολλέ ιδέε ο καθηγητή Ροντρίγκε, τι εκτιμούμε, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά κύριο λόγο να τα σκεφτεί ε, σοβαρότατα. Δεύτερη ερώτηση, κλειδί για την ερχόμενη περίοδο προγραμματισμού. Όντω, εκεί θα έχουμε πολλέ ευκαιρίε να λύσουμε πολλά παρόμοια προβλήματα για τι πολιτικέ για τα αστικά κέντρα. Άρα Εάν μιλάμε για 80% της επικράτειας λαγών, οι στόχοι είναι κοινοί. Τα εργαλεία πρέπει όμως να είναι ποικίλα, διότι είναι διαφορετικό να ε, χαράξουμε πολιτική για αστικά κέντρα, από 80% της επικράτειας, παρόλο που συμμερίζομαι την προτεραιότητα να εργαστούμε επί των αστικών κέντρων, των αδυνατοτήτων των αστικών κέντρων και των ευκαιριών που παρουσιάζουν τις ανάγκες μας. Ευχαριστούμε ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη που δεν μπόρεσα να είμαι από νωρίς και να ακούσω όλους τους ομιλητές. Ο κύριος Ζούμπερ είναι πολύ γνωστός εμπειρογνώμων στην Πολωνία και έχω μια ερώτηση προς αυτόν. Μιλάμε για διάφορα είδη αρεσιμότητας ε, στην πολιτική συνοχή. Ένα από τα πιο έπτυσης και λέτε ότι το σύστημα συγχρηματοδότησης ε, χρησιμοποιείται και πρέπει να χρησιμοποιείται ως κίνητρο. Κάποια κράτη-μέλη ξέρουμε ότι θέλουν τα ποσοστά συγχρηματοδότησης για εξοικονόμηση πόρων. Όμως στη δική σας πρόταση λέτε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε ως κίνητρο. Θα ήθελα να επεκταθείτε πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σομαριζέ τώρα. Ευχαριστούμε θα κληθούμε να διαπραγματευτούμε τον ε, μελλοντικό κανονισμό για τη συνοχή και βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, τις διαπιστώσεις σας και τα ίσως αυτά τα οποία υλοποιήθηκαν για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Λαμβάνω μια νέα προσέγγιση την οποία θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και θα πρέπει να εφαρμόσουμε στην πολιτική συνοχή. Διότι όλο και περισσότερο θα έχουμε αντιμετωπίσουμε, θέλω να πω, αφορά τις ενταφικές ανισότητες. Εμείς ψηφίσαμε να υπάρξει μια, κάτι θέλω να πω, αφορά τις ενταφικές ανισότητες. Εμείς ψηφίσαμε να υπάρξει μια κατεκτές στο Φρανς πράγματι εντυπωσιακό. Και το βλέπουμε παντού στις ανεπτυγμένες αυτές περιφέρειες να έχουμε που είναι το ίδιο ψηλά με αυτά των εξόχων, από απόκεντρων περιοχών που έχουν προβλήματα με την έλλειψη επένδυσεων κτλ. κτλ. Ας δεν ανταποκρίνεται παρκώς σε αυτές. Και ίσως ε, το θέμα των κριτηρίων που έχει ήδη θα πρέπει να μας απασχολήσει ενδελεχώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά όλους γιατί μας δίνετε τροφή για σκέψη και την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ευχαριστώ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλω να σχολιάσω και έχω και κάποιες ερωτήσεις εν συνεχεία. Παγίδα μέσω εισοδήματος στις περιφέρειες. Και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους πέφτουν σε αυτή την παγίδα οι περιφέρειες. Για να μπορέσουμε και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Κάτι διαφορετικό τώρα. Ακούσαμε ότι η πολιτική συνοχή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με την περιφερειακή πολιτική και τις τοπικές πολιτικές. προσοχή στην ε, περιφερειακή διάσταση της ε, πολιτικής συνοχής για να υπάρχει καλύτερη ευθυγράμμιση και συγκρισιμότητα μεταξύ των επιπέδων. Γιατί τα κράτη-μέλη ενίοτε αναπτύσσονται μεν συνολικά, αλλά και συνοχής προς την πολιτική, την περιφερειακή και τις τοπικές πολιτικές. Και τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηστή διακυβέρνηση. Δεν το συζητάμε και πολύ αυτό το θέμα. Είναι όμως μια σημαντική αρχή και πρέπει να εφαρμοστεί. Ίσως θα μπορούσαμε να τονίσουμε να υπάρχει τυπική εφαρμογή και αυτό δημιουργεί και διοικητικό άχθος χωρίς να παρέχει κάποιο πραγματικό όφελος. Υπάρχουν επίσης θέλει και στόχες, άλλο πρόβλημα αυτό θύλακες Γιατί υφίστανται αυτοί οι θύλακε φτώχεια στο εσωτερικό τη. Δεν θα έπρεπε αυτή η περιοχή να μπορεί, αφού έχει πλούτο, να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν παίρνει ενίσχυση, δεν παίρνει υποστήριξη. Εγώ νομίζω ότι τα εσωτερικά τη προβλήματα μια πλούσια περιφέρεια θα έπρεπε να μπορεί να τα λύσει. Επηρεάζει αυτό τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Νομίζω ότι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα φορολογικά συστήματα μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να προσελκύσουν επιχειρήσεις σε κάποιες χώρες ή να προσελκύουν το κέρδος. Ο κύριος Μονσκούρ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ για το πλούσιο περιεχόμενο των παρουσιάσεών τους. Ελπίζω αυτό να μας επιτρέψει να δώσουμε κάποιες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει ένα ζήτημα που επανέρχεται στις παρεμβάσεις. Μιλάμε για απλοποίηση, συνεχώς. Μιλάμε για ευελιξία. Μιλάμε για εμπιστοσύνη και μιλάμε για εδαφικές αποκλίσεις. Παράλληλες αποκλίσεις. Και ο εισηγητής αλλά και τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους αυτό έτσι ώστε να προσπαθήσουμε στα πλαίσια της μελλοντική πολιτικής συνοχή να επιφέρουμε συγκεκριμένε απαντήσεις, διότι αυτό που έχει σημασία για μας σήμερα ε, να ζουν καλύτερα οι κάτοικοι που ζουν εκεί, οι συμπολίτε μα. και ελπίζω όλα αυτά να μας βοηθήσουν να βρούμε απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα εδάφη μας. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητέ, ε, τους ομιλητές ε, για τις παρουσιάσεις. Ήδη έθεσαν πολλά ζητήματα οι συνάδελφοι, οπότε και εγώ θα επικεντρωθώ τονισμό σε οριζόντιο, σε κάθε το επίπεδο, με τις άλλες πολιτικές, μεταξύ των διαφόρων επίπεδων διακυβέρνησης, ε, σε εθνικό, ευρωπαϊκό, τοπικό, περιφερειακό Θα ήθελα να ξέρω να γίνει μια αναφορά στην έξυπνη, στην ευφυή εξειδίκευση, διότι αυτό το συνδέουμε για την ώρα μόνο με τις θεματικές προτεραιότητες, αλλά αυτή η, αρχή της ευφυούς εξειδίκευσης θα μπορούσε να μας βοηθήσει και σε επέδοση συντονισμού μεταξύ της υπαίθρου και των αστικών κέντρων ε, Απευθύνομαι λοιπόν ε, ε, θεωρώ μάλλον ότι αυτό θα πρέπει να αφορά και τους πολίτες, όχι μόνο τις διάφορες, ε, τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, για να μπορούν να προετοιμάζουν καλύτερα τι προτεραιότητες τους και να συζητούν ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε και ποιες είναι οι προτεραιότητες μας βεβαίως. Αυτό είναι το ένα. Και κάτι ακόμα. σε ό,τι αφορά το πώς οι ανάγκες των αστικών κέντρων θα ληφθούν υπόψη. Ναι. Έχουμε εισαγάγει ως πιλωτικό, σε πιλωτικό επίπεδο κάποια εργαλεία που έχουν να κάνουν με τις εδαφικές επενδύσεις. Θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτές τις ε, ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε διαφορετικά το σύνολο της πολιτικής μας και να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή ε, σε αυτό το νέο εργαλείο, σε αυτό το νέο μέσο. Να το ισχύσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόγκοβιτς έχει το λόγο πράστευση Θα επικεντρωθώ στη μετανάστευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα το πρέπει να σταματήσει, διότι θα μας κοστίσει στο μέλλον είτε μιλάμε ε, για Ευρωπαίους από την Ήπεθρο προς τις πόλεις. Υπάρχουν προβολές που μας λένε ότι σε μερικά χρόνια, χρόνια, χρόνια 85% του πληθυσμού θα ζει στις πόλεις. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα. Και θα ήθελα να ξέρω ε, πώς το βλέπετε αυτό στα πλαίσια των προπροσκευαστικών δράσεων, στα πλαίσια της ψηφιοποίησης ε, για την Ήπεθρο. Γνωρίζουμε ότι η ψηφιοποίηση στην Ήπεθρο ε, κέντρων. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε προς την κατεύθυνση αυτή για το μέλλον. Και βεβαίως έχουμε και αυτή τη φιλοδοξία να συνδέσετε αυτές τις πολιτικές ε, καινοτομίες τις οικονομικές πολιτικές με τρεις συνοχή. Και εγώ θέλω, κύριο Σάριμοντ, να ευχαριστήσω τους μιλητές για τις παρεμβάσεις της διαθετικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής που είναι ο έλεγχος. Είπατε ότι υπάρχουν πέντε επίπεδα ελέγχου και ότι είναι υπερβολικό αυτό. Μια συναδελφό σα που είχε έρθει εδώ πριν κάνα δύο μήνε, όταν είχαμε κάνει ένα hearing, από πού ήταν, από την Οβέρνη, δεν θυμάμαι, νομίζω. Και είχε αναφέρει τέτοια πρόβλημα χρόνου. Και ήταν πραγματικά τρελό. Απλό το ερώτημά μου. Τα επίπεδα ελέγχου που εσεί πιστεύετε ότι μπορούμε να καταργήσουμε, ποια είναι. Που δεν χρειάζονται δηλαδή για να γίνει ένας καλός έλεγχος, που αυτός είναι απαραίτητος. Αλλά πια... Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ανέφερα μια-δυο φορές στο πλαίσιο των συζητήσεων για την περιφερειακή πολιτική και προέκυψε και σήμερα το πρωί τις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα φτώχειας εντός συγκεκριμένων περιφερειών. Και όπως υπόθηκε, κρίμα. Αλλά πολλές φορές οι φτωχότερες περιοχές είναι ακριβώς τα κέντρα των πόλεων. Και μάλιστα ευπορότατες πόλεις όπως το Λονδίνο. με τα υψηλότερα ποσοστά παιδική φτώχεια εντό αστικού κέντρου στην, στον Ομένο Βασίλειο. Και αυτό που συμβαίνει στι περιοχέ αυτέ είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα αντίτιμο τη επιτυχία των αστικών πολιτικών για τι ε, αυτές. Υπάρχει ένα φαινόμενο απόκλησης αντί για σύγκληση και δεν είναι κάτι που ισχύει μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ίσως. Υπάρχει ένας, ε, μια συγκέντρωση του πλούτου ε, στις πρωτεύουσες της χώρας. Είναι μεγάλη. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένω να καλυφθεί από την περιφερειακή διακυβέρνηση εντό των περιφερειών. Πάντω αυτό συμβαίνει στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο με περιφερειακού παράγοντε, περιφερειακέ κυβερνήσει να χάνουν, να χάνουν ράξη για τι περιφέρειε του Ηνωμένου Βασιλείου. Ουσιαστικά καταργήθηκε μεγάλο μέρο τη εξουσία του. Δεν πιστεύω ότι απαραίτητο θα πρέπει να είναι ε, ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση εκεί που απέτυχαν οι εθνικέ κυβερνήσει. Όμως πρέπει να δοθεί εδώ η σχετική προσοχή, η δέουσα προσοχή, λόγω και του μεγέθους των αστικών ε, κέντρων και σε σχέση με το μέγεθος κάποιων ε, αστικών κέντρων στην Ευρώπη όπως αυτή που έχει το ΑΕΠ της Αυστρίας και τις διαστάσεις της Δανίας είναι περιοχή, είναι αστικό κέντρο είναι ότι αποτελεσματικότερη από τις επενδύσεις των, της περιφερειακής πολιτικής το είδα και στη δική μου την περιοχή στον Βασίλειο αλλά και αλλού είναι οι επενδύσεις στις υποδομές που επιτρέπουν στην επικοινωνία και τις συγκοινωνίες να αναπτυχθούν. Είναι ότι κάποιες φορές δεν ε, λειτουργεί αυτό σε επίπεδο πόλης αναγκαστικά, αλλά ευρύτερα σε επίπεδο περιοχής, περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν στην περιφερειακή μας πολιτική στο μέλλον να μην ξεχάσουμε ότι θα μας απασχολεί στο θέμα σε αυτές τις περιοχές που διψάνε με αυτές τις τόσο πλούσιες και σκόπιμες παρουσιάσεις σας προκάλεσαν βροχή ερωτήσεων. Θα σας ζητήσω λοιπόν να απαντήσετε ή δυνατόν σε ένα πολύ πρόεδρε. Φοβερά ενδιαφέρον συνολό ρωτήσεων, δεν θα μπορέσω να τις απαντήσω όλες θα επικεντρωθώ σε τρεις βασικούς τομείς. Νομίζω ήταν η βασική πηγή ερωτήσεων. Πρώτα απ' όλα για την παγίδα του μέσου εισοδήματος. Ένα φαινόμενο που πάντοτε υπήρχε. Δεν είναι καινούριο. Μετά η ταξινόμηση και πώς καθορίζει τα αποτελέσματα της συνέπειας της πολιτικής και μετά πιο συγκεκριμένα κάποιες επιλογές για το τι μπορεί να γίνει. Πρώτον, η παγίδα του μέσου εισοδήματος είναι ένα φαινόμενο που δεν είναι καινούργιο, υπήρχε ανέκαθεν, αλλά έχει γίνει πιο ε, διωγγωμένο, διότι από τη μια βλέπουμε η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη και οι οικονομικέ εξελίξει τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε στην Ευρώπη, να επικεντρώνονται κυρίω από τη μια στι πιο δυναμικέ δυνατές πόλεις και περιοχές με το περισσότερο εθνικό κεφάλαιο στην Ευρώπη. Από τα 28 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έλεγα ότι 26 πρωτεύουσες κατά μέσο όρο αναπτύχθηκαν ταχύτερα από ό,τι η υπόλοιπη χώρα. Και με διαφορά είναι πιο δυναμικές περιοχές. Η Ρουμανία τα πάει πολύ καλά, Υπάρχουν αρκετέ αποδείξει που δείχνουν ότι κάποιε χώρε με λιγότερη ανάπτυξη, που ξεκίνησαν από χαμηλά επίπεδα, αναπτύχθηκαν γοργά. Το πρόβλημα είναι κάπου στη μέση και εδώ έχουμε δύο κατηγορίε περιοχών. Από τη μια, περιοχέ που σε πολλέ περιπτώσει έχουν λάβει στήριξη, στήριξη για πολλού λόγου, οι ε, 60-100 χρόνια, ήταν κινητήριε δυνάμει τη ευρωπαϊκή ανάπτυξη και βιομηχανία και τώρα χρειάζονται στήριξη. Είναι ένα φαινόμενο που έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Υπάρχει λοιπόν το θέμα των περιοχών που συγκλίνουν. Έχουμε τη σύγκληση. Περιοχές που επί καιρό ε, είχαν προβλήματα και υποβαθμίστηκαν και περιοχές που κάποια στιγμή είχαν ανθίσει και ήταν πολύ ανεπτυγμένες, τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά παραπέρα και αν δεν τις υποστηρίξουμε δεν μπορούν να συνεχίσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα της ταξινόμησης. Δεν υπάρχει όμως τίποτα εν γενός ε, κακό σε σχέση με την απάντηση. Το έχουμε ετοιμάσει εγώ και ο Μάικλ. Η ταξινόμησή μας ε, είναι απλή. Δεν είναι όμως μόνο το, η ταξινόμηση το πρόβλημα, το τι την κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε εάν έχουν ένα μέρος της χρηματοδότησης, αλλά έχουν και τεράστια εθνική χρηματοδότηση. Διότι το περισσότερο ε, μέρος της εθνικής χρηματοδότησης είναι εδαφικού χαρακτήρα. Δεν υπάρχει εθνική πολιτική που να μην βασίζεται στην εδαφικότητα. Και μάλιστα και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν κολλήσει, βρίσκονται σε τέλμα, σε αδιέξοδο. Έχουν πρόβλημα με το εισόδημά τους και τι έχουν εγκαταλείψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και οι εθνικέ του κυβερνήσει, Και μα το είπε. Ε, δεν είναι μόνο θέμα η αλληλεγγύη εδώ βέβαια. Είναι σημαντική η αλληλεγγύη, αλλά είναι και θέμα ε, του ε, δικού μα του συμφέροντο και τη επιβίωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Με ένα, σε ένα κόσμο ο οποίο είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο ανταγωνιστικό κιόλα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το 80% των περιοχών, αλλά και ένα μεγάλο μέρο σε αυτό το μέσο μέση κατηγορία, Υπάρχουν δύο διαφορετικέ κατηγορίε. Τι είδου μέτρα μπορούμε να προβλέψουμε. Πρώτα απ' όλα διασύνδεση στου θεσμού. Παίρνουμε τι λιγότερο αναπτυγμένε. με το παραδοσιακό μείγμα πολιτικών. Δηλαδή επενδύσει στι υποδομέ, δεξιότητε και να το ματώ, το να κάνουμε τα ίδια και τα ίδια δεν δίνει αποτελέσματα. Είμαι Ισπανός. Θα δώσω παράδειγμα την Πορτογαλία όμω. Βάλτε περισσότερε υποδομέ στην Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν θα υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. <coughs> Αυτέ οι χώρε. Ήδη τα συμπτώματα αυτά αρχίζουν σε κάποια μέρη τη Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιατί ε, οι αδύναμοι θεσμοί ή οι ανεπαρκεί θεσμοί δεν επιτρέπουν να εκμεταλλευτεί κανεί ώστε να αξιοποιήσει το δυναμικό τη επιπλέον επένδυση σε, ε, κοινωνίες, σε υποδομέ συγκοινωνιών. Αλλά και οι επιστροφέ, ε, αυτό το τυπήσουμε, ε, αυτά τα σημεία συμφόρηση στι επενδύσει. Σε πολλέ περιοχέ, όχι μόνο στην Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά αξιότητε στην Πορτογαλία για να μπορέσει ο κόσμος να επιλέξει αν θα μείνει, θα φύγει και αν θα παράγει πλούτο εκεί που βρίσκεται ή όχι. Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση σε επίπεδο δημοτικών, ε, γυμνασίων, λυκείων και χρειάζεται και διαβίου μάθηση. Να μπορέσουν όσοι βρίσκονται σε δυσκολίες ω προ την ε, απασχόληση στην Ιταλία, στη Γερμανία, να αλλάξουν, να ξαναεπινοήσουν το επάγγελμά τους, τη δουλειά τους, να είναι απασχολήσιμοι, ε, προσλήψιμοι σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο ή αλλού, από όπου έρχονται επενδύσεις. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Και εάν ακολουθήσουμε απαράλλακτα τις ίδιες πολιτικές που ακολουθούσαμε στο παρελθόν, οι οποίες λίγο πολύ για μένα υπήρξε μια κάποια αλλαγή στην περιφερειακή πολιτική της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια σε κάποιο βαθμό και ήταν και θετική. Όμως, εάν δεν αλλάξουν ε, οι προποθέσεις της περιφερειακής πολιτικής τα ερχόμενα χρόνια δεν θα αλλάξουν και πολλά. Είναι λες και ε, προσπαθούμε να βάλουμε χρήμα αντιμετωπίζοντα ακριβώ τι ίδιε πηγέ προβλημάτων χωρί να πετυχαίνουμε αποτελέσματα. Αυτό που θέλουμε είναι να επενδύσουμε χρήματα για τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή την ευημερία των ανθρώπων που ζουν σε συγκεκριμένο είδο περιοχών που έχουν στην Ευρώπη. Σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε πολύ πιο δυνατά και περισσότερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να εστιάσω σε ορισμένα από τα στήματα που τέθηκαν. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι αρκετές παρατηρήσεις αφορούσαν τις κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στις αστικές περιοχές. Και έτσι μου δίνεται και μια δυνατότητα να επισημάνω ότι οι κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις στις αστικές περιοχές είναι και οι πολυπλοκότερες, μακράν. Και η πολιτική συνοχή έχει την έντονη τάση να επενδύσει σε υποδομές. Όμως η κοινωνικο οικονομική διάσταση ότι είναι πιο πολύπλοκη. Χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από την πολιτική συνοχή. Και πρέπει να δούμε τη μετατόπιση ε, της χρηματοδότησης ως ενδεχόμενο για την αντιμετώπιση αυτών των ε, κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων που επηρεάζουν τον κοινωνικό ιστό σε σχέση με δύο θέματα που αναφέρθηκαν, μετανάστευση και φτώχεια. Εγώ βέβαια θα προτιμούσα να γίνεται λόγος για μετανάστευση ή καλύτερα κινητικότητα τόσο εντός Ένωσης αναφέρθηκε νομίζω κινητικότητα του εργατικού δυναμικού από τις χώρες του Νότου στην Βορειοανατολική στη βορειοδυτική Ευρώπη και από την Ανατολή προς Η κινητικότητα φυσικά και εξηγείται λόγω των εδαφικών ανισοτήτων. Αν δεν υπήρχαν δουλειές, οι περισσότερες δουλειές ε, στην περίοδο της κρίσης σε άλλες χώρες και αν υπήρχαν αυτές οι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία δεν θα φεύγανε οι νέοι αυτών των χωρών να πάνε σε άλλες χώρες να εργαστούν. Φυσικά και υπάρχει το πρόβλημα. Το θέμα είναι η κινητικότητα να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να βελτιώσει και τις δεξιότητες στις ίδιες τις περιφέρειες. Κάτι άλλο που βλέπουμε και το είπαν και ορισμένοι ε, ευρωβουλευτές είναι το εξής. Και είναι ενδιαφέρον. Ότι υπάρχουν θύλακες φτώχειας στις αστικές περιοχές και η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Η 7 για τη συνοχή δείχνει ότι στις 15 χώρες μέλη παλαιότερες τα επίπεδα φτώχειας είναι υψηλότερα σήμερα από ό,τι πριν τη χρηματοπιστωτική κρίση. Και στις 13 νέες κάπως έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Δηλαδή, η θύλα και στόχια συστιάζουν κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Βέβαια και στις πόλεις αυξάνονται τα ποσοστά φτώχειας. Στις 15 χώρες η κατάσταση αυτή έχει να κάνει και με το γεγονός ότι πάντοτε υπήρχαν φυλακιστώ στόχοι στις πόλεις. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ότι πάντοτε υπήρχαν θηλυκές στόχοι στις πόλεις. Και αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Ο συνάδελφος από τον Ηνωμένο Βασίλειο μίλησε και για την ε, παρενέργεια, μπορώ να το πω έτσι, της οικονομικής επιτυχίας των αστικών περιοχών στις πρωτεύουσες και το βλέπουμε αυτό, ότι αναπτύσσονται στην Ευρώπη, αλλά αυτό επηρεάζει παράπλευρα τα επίπεδα φτώχειας. Ιστορικά δε προσελκύει μετανάστες ε, η πρωτεύουσα. Πρόσφυγες και μετανάστες κυρίως στις αστικές πηγαίνουν, ε, στις μεγάλες περιοχές. η προσέγγιση πρέπει να στηρίζεται και στο μέρος και στον άνθρωπο. Και εκεί που εστιάζω, εκεί που υπάρχει συγκεντρωμένη φτώχεια, εκεί πρέπει να γίνουν και οι κατάλληλες υποδομές. Κοινοοικονομικές προκλήσεις λοιπόν. Για την αντιμετώπιση χρειάζεται συνέργεια μεταξύ των κονδυλίων των διαφόρων ταμείων. και είναι πολυεπίπεδα τα προβλήματα, πολύπλοκα. Χρειάζεται λοιπόν διατομεακή εγκάρσια προσέγγιση. Διάφορες ε, πολιτικές πρέπει να συμμετάσχουν γιατί υπάρχουν παραδείγματος χάρη ζητήματα υγείας, έλλειψης κινητικότητας, ανεργίας. Ε, άκρος πολύπλοκα θέματα. Και ανεργία δεύτερης γενιάς μάλιστα. ITIs μπορούν να βοηθήσουν, το είδαμε στην Πολωνία, αλλά σε άλλες χώρες δεν χρησιμοποιούνται λόγω της ε, γραφειοκρατικής πολυπλοκότητας. Ε, νομίζω η Γερμανία είναι ένα παράδειγμα. Καλό είναι να δούμε λοιπόν τα ITIs αυτά πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Απλούστευση τώρα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να εστιάσω σε δύο θέματα. Το πρώτο φαίνεται τεχνικό, αλλά δεν είναι. Μιλάω για τη συγχρηματοδότηση. Το σύστημα συγχρηματοδότηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο. Τελικά, πάντοτε ε, για χρήματα και προπολογισμό θα συζητάμε. Αυτό που εννοούσα εγώ όμω είναι να μην συστάμε τώρα αυτή τη στιγμή για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης, αλλά να οργανώσουμε το σύστημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συγχρηματοδότηση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για την υποστήριξη των πολιτικών αυτών που θέλουμε να ενταχθούν στη νέα πολιτική συνοχή. Τι θέλω να πω με αυτό. Μιλάμε για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, επί παραδείγματι. Και εδώ ακούσαμε ότι υπάρχουν δυσκολίες με το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Κοινωνικό Ταμείο. Πώ συνεργάζονται αυτά τα δύο μεταξύ του. Πρέπει να οργανώσουμε κατά τέτοιο τρόπο το σύστημα ώστε όταν κατατεθούν έργα, project τα οποία μπορούν να συνδυάσουν κοινωνικό ταμείο και περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό είναι πολύ καλό. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να γίνει και να ειδωθεί και στο πλαίσιο αυτό που ανέφερα. Μιας νέας δέσμη μέτρων δηλαδή, για όλα αυτά τα εργαλεία. Και εκεί θα το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Σε αυτά τα συνδυασμένα project μπορούμε να έχουμε χαμηλότερα ποσοστά συνδυασμένα. Και αυτό είναι κίνητρο να καταθέσει κάποιο τέτοια project. Δηλαδή, να μην απομονώνουμε Φτιάχνω δρόμους, ένα project, δεύτερο project, στηρίζω το ανθρώπινο κεφάλι, την Στην Πολωνία σίγουρα ε, τα προγράμματα αποδίδουν, δίνουν νέε δεξιότητε, αλλά βρίσκουν θέσει δουλειά τα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν βρίσκουν και τι κάνουν, όπω είπατε, μεταναστεύουν. Έχουμε αποτελεσματική κοινωνική πολιτική που χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, τελικά όμω οι περιφέρειες δεν ωφελούνται παρότι εκεί ε, δουλεύει το ΕΚΤ. Γιατί φεύγει ο κόσμος. ITIs. Είπατε να είναι σημαντικά. Γιατί να μην δώσουμε κίνητρα για συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών. Με συμμετοχή ιδιωτικών και δημόσιων εταίρων. Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο. Ένα τέτοιο σύστημα συνεργασίας, όχι μόνο μεταξύ των δημοσίων αρχών, αλλά με την παρουσία και άλλων εταίρων πάλι η συγχρηματοδότηση θα είναι λιγότερη ή περισσότερη, ανάλογα με το πώς το βλέπει κανείς το πράγμα. Και το τρίτο πολύ απλό παράδειγμα είναι ότι έχουν διαφορετικούς κανόνες για την πολιτική συνοχή και για το ΕΦΣΙ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι κρατικέ ενισχύσει. Θέλουμε να έχουμε παραγωγικού τομεί. Αν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υπάρχουν πολλά έργα, project στην πολιτική συνοχή που έχουν ευρωπαϊκή προστεμένη αξία στου παραγωγικού κλάδου, τότε γιατί έχουμε κανόνε για τι κρατικέ ενισχύσει. Ε, μας αρέσει η έννοια αυτή σε όλους. Και σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο έχουμε εκπονήσει στρατηγικές όμως, από ό,τι προκύπτει, δεν αρκεί αυτό η εκπόνηση ωραίων στρατηγικών. Πρέπει να εφαρμόζονται αυτέ οι στρατηγικέ και να είναι και διαχειριστικό εργαλείο, όχι σημείο αναφορά απλά που λέω ότι ορίστε να έχουμε στρατηγική. Πρέπει να έχει απτά αποτελέσματα. Να οργανώνει το σύστημα. Σε αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ. Πρώτα για το ΕΚΤ αλλά και την ε, ελάφρυνση των ελέγχων. Τώρα, τα αποδεικτικά στοιχεία, η δίκαια, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί τόσο καλά και βεβαίως ε, λάβετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία αν θέλετε. Σε κύριο Ζουλό, στον κύριο για τις ανησυχίες που έχουμε για το ΕΚΤ, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ε, αυτό, λάβετε αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία αν θέλετε. Σε κύριο Ζουλό, στον κύριο για τις ανησυχίες που έχουμε για το ΕΚΤ, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, αυτό το διαφορετικό ταμείο για την περιφέρεια Ile-de-France είναι κεφαλαίου σημασίας. Ε, είναι η μόνη περιφέρεια της Γαλλίας όπου το ε, κοινωνικό ταμείο ε, είναι υψηλότερο από το Φέντερ και βεβαίως αυτό σχετίζεται με πολύ συγκεκριμένες προβληματικές που αφορούν την περιφέρειά μας ε, εντός της περιφέρειας κάτι που δεν ελέγχθη σήμερα το πρωί για έναν απλό λόγο. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο των μικρών δομών, ιδιαίτερα των μικρών ε, συλλόγων ε, που δεν χρειάζονται δάνειο, δεν χρειάζονται κάποια εγγύηση για να δανειοδοτηθούν σε συγκεκριμένες θεματικές. Και να ε, ε, ελαφρύνουμε κάπως τα κριτήρια του πλαισίου, γιατί δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το πλαίσιο απόδοσης είναι σημαντικό λοιπόν να το δούμε και αυτό. Και να απαντήσω τέλος ε, τα ευρωπαϊκά επίσης σώματα ε, ελέγχου δεν βεβαίως δεν και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο στις περιφέρειες τουλάχιστον στα εθνικά εδάφια όπου υπάρχουν περιφέρειες ε, στις αρχές προσπάθεια έγινε αυτή η δουλειά και τώρα νομίζω πως είναι λογικό και νομίζω περισσότερο ή λιγότερο και να υπάρχει ένα επίπεδο ελέγχου ευρωπαϊκό. Λογικό και αυτό, μια και πρόκειται για χρηματοδότηση, για χρήματα ε, ευρωπαϊκής προέλευσης. Αυτή είναι η δύο προσανατολισμοί. Τώρα, πέρα από την απλοποίηση, νομίζω πως αυτό που είναι πολύ σημαντικό και βεβαίως πάει πέρα από την πολιτική συνοχής, είναι να δώσουμε ένα νόημα και μια συνοχή, ε, μια συνέπεια. Ε, εάν ε, οι διαδικασίες, οι λεπτομέρειες εφαρμογής έχουν διάποτε και αυτές από την ίδια συνέπεια, τότε υπάρχει και ένα κίνητρο περισσότερο, υπάρχει μια μόχλευση και αντιλαμβάνεται, αντιλαμβάνεται και η δοχή. Όχι το να έρθουμε, ευχαριστούμε όλους τους ομιλητές και για το πολύ ενδιαφέρον αυτό εργαστήρι. Και τώρα περνάμε στο επόμενο. Ναι, θα είμαι σύντομος. Είμαι ο Λούις Ντέξτρα, είμαι ο εκδότη αυτή τη εκθεση για τη συνοχή. Άκουσα μεγάλη ενδιαφέρον αυτή τη συζήτηση. Το θέμα και επισημαίνεται και στην έκθεση περί συνοχής, αλλά θέλω να εξηγήσω δύο πράγματα περί αυτού. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι διαφορά μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών τη υπαίθρου. Σε καμία περίπτωση. Οι πόλεις, σε αυτέ τι περιοχέ του μέσου εισοδήματο. Μερικές θα πάνε κάπως καλούτσικα, αλλά όχι αρκετά, για τις μεταξύ πόλεων και περιοχών τη υπαίθρου. Επίσης, να πω ότι για την παγίδα του μέσου εισοδήματο θεωρούμε ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια ε, διαδικασία ομαλή εύρυθμη, αλλά με, πολλές, ε, με πολλούς τριγμούς, ε, με πολλές αναταράξεις, πρόσβαση στις πιστώσεις, τα δάνεια. Πολλές από τις περιοχές λοιπόν του μέσου εισοδήματος απαιτούν πολύ περισσότερο ολοκληρωμένη, συντονισμένη προσέγγιση για να μπορέσουν να περάσουν σε καινοτομότερε και ψηλότερη παραγωγή. προσφερθούν στις περιοχές μέσω εισοδήματος για να κάνουν το άλμα ποιότητας που περιμένουμε. Ως προς τις πόλεις, Πολλές από αυτές είναι κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, κάποιες όχι. Έχουμε πόλεις με οικονομία σημαντική, κάποιες που συρρικρώνονται πληθυσμιακά και ακόμη και πιο επιτυχείς περιλαμβάνουν φοβερούς θύλακες φτώχειας. Όλα αυτά ε, ως προς την εδαφική διάσταση. Προσπαθούμε να την ε, διοργανώσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Στο παρελθόν άκουσα υποστηρικτικά σχόλια αλλά και επικριτικά για το πόσο περίπλοκο είναι όλο αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε σε δύο επίπεδα, ανάλογα με το τι μέλλον θέλουμε να προσφέρουμε, να υπάρχει ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, η πολιτική να επικεντρώνεται εκεί που μετράει και οι πολιτικές να προσαρμόζονται στις ε, ανάγκες και το δυναμικό της κάθε περιοχής. Συμφωνώ με τον κύριο Ζούμπερ ότι μιλάμε για μια πολύ ε, λεπτότερη διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ των ε, διαφόρων περιοχών και εντός των των ίδιων περιοχών ανάλογα με τους διάφορους φύλακες. Μια πιο διαφοροποιημένη λοιπόν προσέγγιση για τις διάφορες περιοχές και όχι μικροδιαχείριση αλλά ευελιξία για τα κατημέλη ώστε να μπορούν να στοχεύσουν τις περιοχές που θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν οι περισσότερη στόχευση. Το τελευταίο που θα πω είναι για το management και το σύστημα ελέγχου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο κόσμο το σημείωσε αυτό και αντί να πει απλώ απλούστευση, κάτι που το επιδιώκουμε εδώ και 20 χρόνια, ε, περάσαμε στην ριζοσπαστική απλούστευση. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέτετε για να σας παρουσιάσω την ε, γνωμοδότηση αυτή Είμαι αντιδήμαρχος στην... Ε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε να ζητήσω από όσους ε, φεύγουν τώρα να το κάνουν αυτό σιωπηρά. Και ησύχως διότι δουλεύουμε ακόμα. Ε, είμαι λοιπόν υπεύθυνο για θέματα δημοτική συνεργασία, αλλά και ο ίδιο ανήκω σε δημοτικό συμβούλιο. Να σα δείξω τώρα από πού έρχομαι. Βόρειο μέρο τη Δημοκρατία τη Τσεχία. Αυτό βλέπουμε. Ε, έχουμε ένα μέρο επίση ε, τη Πολωνία και τη Ανατολική Γερμανία. Ένα μέρο με πολύ δύσκολη ιστορία. Προσαρτήθηκε και είχαμε και κατοχή από τη Γερμανική Αυτοκρατορία πριν από τον πόλεμο ήδη αλλά και μετά τον πόλεμο όλοι οι Γερμανοί ε, κάτοικοι που ζούσαν εκεί από αιώνε παραδοσιακά ε, απελάθηκαν, ε, ανταλλάχθηκαν οι πληθυσμοί και ήρθαν νέοι κάτοικοι να μείνουν εδώ. Τι σημασία έχει αυτό, γιατί τα προγράμματα ακριβώ από πολίτη σε πολίτη έχουν βοηθήσει να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Να σας δώσω τώρα ένα παράδειγμα προγράμματος. Ο Ιωπέρα, ε, η Ορχήστρα των Νέων, διευθυντές μουσικών σχολών οδείων και από τι τρει χώρε συγκεντρώνουν τους καλύτερους μαθητές τους σε μία ορχήστρα. Κάθε καλοκαίρι σε μια κατασκήνωση εξασκούνται όλοι μαζί κάνουν πρόβες ε, και μετά οργανώνουν και ένα κονσέρτο. Εάν έβλεπε κανεί μια τέτοια συναυλία, θα έβλεπε τι ωραίο κλίμα επικρατεί. Διότι υπάρχουν παιδιά από τρει χώρε που καμιά φορά δεν γνωρίζουν καν ε, τη γλώσσα των ΔΕ αλλά συνεννοούνται μέσω τη μουσική που είναι μια άλλη πολύ δυνατή γλώσσα και πολύ δυνατό εργαλείο. Πολύ σύντομα λοιπόν να τονίσω ότι στι γνωμοδότε μα προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε την προστιθέμενη αξία αυτού του προγράμματο. Διότι είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλο τη διασυνοριακή συνεργασία. Θα έπρεπε μάλλον να είναι, δεν είναι ακόμα. Κάποιε φορέ μπορέσαμε να αναπτύξουμε ευρύτερα προγράμματα. Τα Προγράμματα θα μπορούσε κανεί να πει ότι λειτουργούν ω εκολαπτήρια για τη μελλοντική μα συνεργασία. Δηλαδή ένα λεξικό για αστυνόμους λόγου χάρη, ένα γλωσσάρι, για να μπορούν να διεξαγάγουν κοινού να διεξάγουν κοινού ελέγχου και να έχουν αποτελεσματικότερη συνεργασία στο μέλλον, σε σημεία ελέγχου στα σύνορα, λόγου χάρη ή κοιτάξαμε να διευκολύνουμε την ε, εκπαίδευση και την εξοικείωση με την κουλτούρα των γειτονικών χωρών. Θέατρο, την εξοικείωση με την κουλτούρα των γειτονικών χωρών. Θέατρο. Έχουμε ε, διευκολύνει τις διαπροσωπικές επαφές με ισχυρές εταιρικές σχέσεις και με συμμετοχεύουν ε, την κοινωνία των πολιτών. Δεν αφορούν φορεί, κρατικού φορεί, ε, κυβερνήσει, υπουργεία, αλλά την κοινωνία των πολιτών. Συνήθω μιλάμε για αθλητικού συλλόγου, νηπιαγωγία, σχολεία, ε, συλλόγου ορειβατών. Αυτοί ε, είναι τα μέλη των προγραμμάτων αυτή Όταν όμως στοχεύει αυτές τις συγκεκριμένες ε, πιο περιορισμένες περιοχές μπορεί να στοχεύσει και τοπικά προβλήματα, τοπικά ζητήματα που έχουν ε, σημασία για την καθημερινότητα. Και τα τελευταία δύο σημεία που ήθελα να αναπτύξω είναι η προστεθεμένη αξία των προγραμμάτων αυτών. η ενίσχυση της εμπιστοσύνης. 25 χρόνια επέτειος Γιορτάσαμε 25 ετή επέτειο ε, πριν από λίγο καιρό και αν θυμάστε στην τούρτα που κόψαμε το τελευταίο στρώμα ήταν η εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το θεμέλιο όλων. Αυτή είναι η προστιθέμενη αξία των ε, διαφόρων ε, προγραμμάτων που σας παρουσίασα και τώρα πολύ σύντομα να θίξω το θέμα του αποκεντρωμένου management της διαχείρισης. Τα προγράμματα αυτά από πολίτη σε πολίτη, τέλος πάντων ε, μικρής κλίμακας στην ουσία, δεν υπάρχουν παντού. Το 1 τρίτο είναι προγράμματα συνεργασία, αλλά είναι μέρο άλλων μεγαλύτερων προγραμμάτων κάποιε φορέ. Και όπου υπάρχουν, έχουν ένα μικρό ποσοστό ε, κονδυλίου από το μεγαλύτερο κονδύλιο του προγράμματο, το οποίο αποκεντρωμένα ε, αποστέλλεται σε συγκεκριμένε περιφέρειες ή διασυνοριακέ δομέ. Κάποιες φορές μιλάμε για 2%, κάποιες φορές κατ' 20%. Συνήθως είναι 5-10% της συνολικής ποσόστοσης του προγράμματος. Το παίρνει λοιπόν η μικρότερη αυτή περιοχή, λόγω χάρη για τα σύνορα Τσεχίας-Πολωνίας, που είναι 350 χιλιόμετρα μόνο, έχουμε έξι μικρούτσικα ε, προγραμματάκια που διατίθενται στους ε, μικρούς ετούντες. Οι περιοχές κάποιες φορές επίσης με ένα συνολικότερο πρόγραμμα παίρνουν όλο το κοντήλι και το διαιρούν στα μικρότερα μικρούτσικα προγραμματάκια. Οι δομές λοιπόν αυτές όπως ε, σε ποιον θέλουν συνεργασία για ποιο σκοπό κάνουν την ερμηνεία του προγράμματος και των κανόνων του, φέρουν τους ανθρώπους σε επαφή, τους εξοικειώνουν μεταξύ τους, τους συνεργάτες. Δεν είναι απλώς λοιπόν μια διαχείριση από μακριά. Προστιθέ πρόγραμμα στην Πολωνία πρέπει να ταξιδέψουν 3,5 ώρες στο, στη γραμματεία του Υπουργείου για να μπορέσω να υποβάλω την αίτησή μου. Για μένα όμω, στη δική μου την περιοχή, για αυτό το μικρό προγραμματάκι, μπορώ να είμαι εκεί μέσα σε ένα τεταρτάκι. Και γεωγραφικό είναι πολύ πιο απλό. Αλλά τα προγράμματα είναι πολύ απλούστερη. Μια ετησούλα, μια σφραγίδα και το κονδύλι εκταμιεύεται. Ουσιαστικά το πρόγραμμα ανοίγει σε μεγαλύτερο αριθμό ετούντων από μικρές δημοτικές αρχές μέχρι με κυβερνητικές οργανώσεις και για την πολιτική συνοχή και τη διασυνοριακή συνεργασία με τα σχετικά προγράμματα μετά το 2020. Ξέρω ότι εδώ συζητούμε το 5-10% του 3% που αποδίδεται στην διασυνοριακή συνεργασία από το Σύνολο της της Πολιτικής Συνοχής. Είναι ένα πολύ μικρό ποσό. Όμως μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Να ε, διασφαλίζονται και από τους κανόνες και τους κανονισμούς. Για την ώρα δεν συμβαίνει αυτό. Οι μικρό, μεγαλύτερες περιοχές που συνεργάζονται με την Επιτροπή από μόνο του παίρνουν την πρωτοβουλία και δημιουργούν αυτά τα κονδύλια για τα μικρότερα προγράμματα, αλλά καλό θα ήταν να υπάρχουν και στον κανονισμό, να είμαστε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει σχετική ζήτηση, ε, εφόσον υπάρχει μάλλον σχετική ζήτηση. Εάν όχι, δεν χρειάζεται. Πάντω θέλουμε σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο να είναι μέρο του προγράμματο αυτά τα προγράμματα. Επίση με αποκεντρωμένη διαχείριση. Αυτό θέλουμε να διατηρηθεί. Η... Και τα προγράμματα αυτά θέλουμε να παραμένουν όσο δυνατόν απλούστερα. Με την απλούστευση της διαδικασίας κόστου. Η τελευταία φράση τη νομοδότηση τώρα και η τελευταία μου διαφάνεια. Τι θέλουμε να πετύχουμε και σα ευχαριστώ πολύ. Προσπάθησα να είμαι στο το δυνατόν πιο συνοπτικό στην παρουσίασή μου, αλλά ελπίζω ότι σα τα εξήγησα καλά και έδωσα αρκετέ αφορμέ για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ για αυτή την παρουσίαση. Αυτά τα μικρή κλίμακα project ε, είναι στο πλαίσιο του Interreg. Αλλά είναι κάπως διαφορετική διαχείριση. Είναι πιο εύκολο, όπως είπατε, είναι πιο κοντά στους πολίτες, ε, δυνητικούς δικαιούχους. Υπάρχουν πολλά εμπόδια για την υλοποίηση σε σχέση με τη δίκηση και τη διοικητική ικανότητα. Στο ίντερεκ να μεταφερθεί η εμπειρία των ευρωπεριφερειών και της διαχείρισης αυτών των μικρής κλίμακας προγραμμάτων. Θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει κάποια σημεία. για την παρουσίαση αυτή. Διότι αυτά τα project για τον άνθρωπο ε, είναι μικρής κλίμακας, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικά και έχουν πραγματικά προστιθέμενη αξία. Σε πολλές περιπτώσεις με αυτά τα μικρά project, όπως είπατε και ξεκινώντας την παρουσίασή σας, το ερώτημά μου λοιπόν είναι, ή μάλλον να πω και κάτι ακόμη, γνωρίζουμε ότι η χρηματοδότηση για το Interreg είναι πολύ περιορισμένη. Η χρηματοδότηση δεν για τα μικρά πρωτό να ζητήσουμε αύξηση της χρηματοδότησης του Ίντερεγ και της διασυνορικής συνεργασίας εν γέννη στο πλαίσιο της περιφερειακής και διατομιακής συνεργασίας. Απάντηση. Η προσωπική μου άποψη και η άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών είναι ότι ναι, πράγματι έχετε δίκιο. Αν διαβάσει κανείς ε, το έγγραφο προβληματισμού για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γνώμονας θα έπρεπε να είναι ακριβώς αυτός. Για το πώς... Αν διαβάσει κανείς ε, το έγγραφο προβληματισμού για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο γνώμονας θα έπρεπε να είναι ακριβώς αυτός για το πώς δαπανώνται τα χρήματα το Εράσμους είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Ότι δηλαδή έχουμε... Μιλήσαμε για τη συνοχή, σύντος μιλάμε για το ΑΕΠ. Ας πάμε τη συζήτηση κάπου αλλού τώρα, στην ποιότητα ζωής για παράδειγμα. Για να υπάρχει ποιότητα ζωής είναι πολύ σημαντικό να έχεις καλούς γείτονες. Αν έχεις κακό γείτονα, μπορεί να είναι η ζωή σου κόλαση. Ενώ αν έχεις έναν και μετά να είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο με πολύ καλή απόδοση αυτή τη επένδυση. Κάποιε φορέ δεν βλέπουμε αυτά αποτελέσματα όπω με τα μεγάλα project. Δηλαδή δεν έχουμε αύξηση τη χρηματοδότηση τη διασυνορικής συνεργασία. Αυτό σημαίνει περισσότερα χρήματα και για αυτά τα μικρή κλίμακα σχέδια από τον άνθρωπο στον άνθρωπο και με την αξία που έχουν αυτά τα μικρή κλίμακα έργα. Είπα ότι είναι κολαπτήρια για μεγάλα project. Εγώ εδώ και 25 χρόνια εργά με αυτούς που εφαρμόζουν το project στην πράξη και αν υπάρχει καλή συνεργασία μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Αν δεν υπάρχει αυτή η βασική εμπιστοσύνη είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τον άλλο, τα σύστηματα διαχείρισης που μπορεί να ήταν διαφορετικά τα έμαθαν ε, και μετά κατέθεσαν μια μακροχρόνια εμπειρία. Για τη διασυνορική συνεργασία και το τι γίνεται γενικότερα με το ίντερνετ τα αποτελέσματα δείχνουν το αντίθετο. Υπάρχει μια αντίφαση με αυτά που μας λέτε εσείς, ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο Interreg. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι διαφορετικό. Τόσα πολλά τα μικρά τα προγράμματα και τόσα πολλά τα τέψουμε τη διοικητική, τη διγραφειοκρατική δομή για να είναι αποτελεσματικότερες οι σχέσεις συνεργασίας